le monde. Euh, je vous propose qu'on puisse euh, débuter notre réunion. Ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Οι διερμηνείς έχουν να κάνουν μια ανακοίνωση. Ε, η εργασιακή διάνεξη ανάμεσα στους διερμηνείς και την διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βρίσκεται στην τρίτη εβδομάδα. Παρ' όλα αυτά η διοίκηση δεν έχει έρθει ακόμα σε επαφή μαζί μα για να δοθεί μια λύση. Πολλέ μάλιστα καμπίνες έχουν επιστρατευθεί. Ε, Ω αλληλεγγύη προ αυτέ τι καμπίνε και για να μην γίνονται διακρίσει εναντίον βουλευτών και γλωσσών, η ελληνική καμπίνα αποφάσισε να αναστείλει την στάση εργασία που είχε προγραμματιστεί για σήμερα. Παρ' όλα αυτά, δεν θα εργαστούμε πέραν του προγραμματισμένου χρόνου εργασία. Ευχαριστώ. Je vous remercie. Ας ξεκινήσουμε την απογευματινή μας συνεδρίαση με μια ακρόαση για την ενίσχυση των δεσμών εμπορική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Λατινικής Αμερικής. Ο πρόεδρος Λάγκε δυστυχώς δεν μπορεί να παραστεί αυτή τη στιγμή, θα έρθει μάλλον αργότερα να ευχαριστήσω το Διπλωματικό Σώμα και του πρέσβει που είναι παρόντες, καθώ επίση και του εμπειρογνώμονε ε, που θα μοιραστούν μαζί μα τη γνώση του για το θέμα. Όπω γνωρίζετε, κατά τη διάρκεια τη θητεία μα έχουμε εργαστεί σκληρά για να ενισχύσουμε του δεσμού με τις χώρες τη Αμερική, εφαρμογή συμφωνιών με την Κολομβία, τον Ισημερινό και το Περού, καθώς επίσης και με την Κεντρική Αμερική, διαπραγματεύσει με τη Χίλη και το Μεξικό για τον εξυγχρονισμό των συμφωνιών και οι εμπορικέ διαπραγματεύσουμε την Μερκοσούρ είναι σημαντικά θέματα της εργασίας μας. Έχουμε καλέσει πολλούς αρκετούς εμπειρογνώμονες και θεσμικούς εκπροσώπους για να εμβαθύνουμε στο θέμα αυτό. Το πρώτο πάνελ θα μιλήσει για τις ε, τρέχουσες διαπραγματεύσεις, ενώ το δεύτερο για την εφαρμογή των υπαρχουσών ε, συμφωνιών. Ε, εξυγχρονισμό των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων με τη Λατινική Αμερική είναι το θέμα του πρώτου πάνελ. Δίνω το λόγο στην κυρία Χρεντά, ε, εκτελεστική διευθύντρια για τις ε, χώρες της Αμερικής στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Σχέσεων. Thank you very much, madam. Thank you very much for... Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Όπως είπατε και εσείς, ε, αυτή τη στιγμή ε, διαπραγματευόμαστε τον εξυγχρονισμό ορισμένων συμφωνιών με τις λατινοαμερικανικές χώρες, πιο συγκεκριμένα τρεις. Περιλαμβάνουν και πολιτική ε, συνεργασία και εμπορικό κομμάτι αυτές τις συμφωνίες. Τρεις, διαπρα... τρεις συμφωνίες διαπραγματευόμαστε, όπως σας είπα. Καταρχήν με το Μεξικό, ε, διαπραγματεύσεις που έχουν προχωρήσει πολύ. Βρισκόμαστε στα τελευταία στάδια. Έχουμε κλείσει το θέμα της πολιτικής συνεργασίας από τον Νοέμβρη και όπως γνωρίζετε συμφωνήσαμε επί της αρχής και για το εμπορικό κομμάτι στο τέλος Απριλίου. Οπότε τα εκκρεμή θέματα αφορούν τεχνικά ζητήματα τα οποία θα ολοκληρώσουμε ε, σύντομα. Πολύ σύντομα μάλιστα θα περάσουμε στη μετάφραση των κειμένων. Αυτή η συμφωνία είναι από τις πιο σύγχρονες και επίκαιρες που έχουμε με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής και της Καρεβικής. Το Μεξικό ήταν ο πρώτος εταίρος με τον οποίο ξεκινήσαμε διαπραγματεύσεις ε, πολλά χρόνια πριν, το 1997. Τότε ε, αυτή η συμφωνία και είναι και στρατηγικός μας εταίρος. Αυτό το απηχεί η συμφωνία. Γι' αυτό έχουμε και πολλά καινούργια κεφάλαια, επικαιροποιημένα, και οι συνεργασίε επενδύσει επίση είναι κάτι πολύ καινούριο. Οι συνάδελφοι από τη Γενική Διεύθυνση ε, Trade ε, θα συμπληρώσουν. Ο πολιτικός διάλογος με το Μεξικό είναι πολύ στενός. Αντιμετωπίζουμε θέματα παγκόσμιας, ε, παγκόσμιου ελληνικού όπως ενέργεια, κλιματική αλλαγή, περιβάλλον, ψηφιακή οικονομία, βιώσιμη ανάπτυξη, μακροοικονομικές πολιτικές προφανώς, ε, που θα πρέπει να δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για τις επιχειρήσεις μας και έχουμε και πολύ καλά αποτελέσματα στην έρευνα, την ανάπτυξη, ιδιαίτερα στον τομέα της ε, πληροφορίας και τεχνολογίας, IT. Η δεύτερη συμφωνία, την οποία μόλις ξεκινήσαμε να διαπραγματευόμαστε πριν από μερικούς μήνες, είναι η συμφωνία με την Χιλή. Εκεί η κατάσταση έχει αλλάξει γιατί είχαμε αλλαγή στην κυβέρνηση της Χιλής. Ακόμα όμως και εδώ έχουμε δει πολύ γρήγορη και σημαντική πρόοδο ε, και εδώ έχουμε μια ε, ευρεία σφαιρική συμφωνία που περιλαμβάνει πολιτική συνεργασία και έχει και ένα εμπορικό κομμάτι. Τρεις γύρια διαπραγματεύσεων έχουν ήδη ολοκληρωθεί για το εμπόριο και στον επόμενο γύρο θα ξεκινήσουμε αύριο και να συζητάμε το θέμα της πολιτικής συνεργασίας και εδώ έχουμε πολλές προσδοκίες. Η Γενική Διεύθυνση Trade το Μάιο ξεκίνησε μία μελέτη, ε, ε, ε, μελέτη αντικτύπου ε, καθώς επίσης και διαβούλευση μέσω του διαδικτύου για να πάρουμε τα σχόλια των επιχείρησεών μας και των διαφόρων ευρωπαϊκών φορέων. Αυτή τη στιγμή ε, είμαστε, όπως σας είπα, στον τρίτο γύρο για για το εμπόριο. Έχουμε προχωρήσει σχετικά καλά. Ε, δεν έχουμε πάει πολύ μακριά ακόμα, είναι νωρί. Ε, έχουμε πολλές φιλοδοξίες, διότι η καινούργια κυβέρνηση στη Χιλή δήλωσε ότι επιθυμεί διακαώς να ολοκληρωθούν σύντομα οι διαπραγματεύσεις. Οπότε ελπίζουμε ότι θα φτάσουμε σε μια πολιτική συμφωνία πριν το τέλος του χρόνου. Τρίτη διαπραγμάτευση, την οποία βλέπετε συχνά στον τύπο, είναι η διαπραγμάτευση με τις χώρες του Μερκοσούρ. Είναι περίπλοκη, Ε, η ο τελευταίος γύρος διαπραγματεύσεων έλαβε χώρα 6 με 8 Ιουνίου στο ε, Μοντεβιδέο. Ελπίζουμε ότι θα καταλήξουμε σε πολιτική συμφωνία. Ε, έχουμε κλείσει το θέμα της πολιτικής συνεργασίας. Το εμπορικό σκέλος ακόμα όμως εκκρεμεί για τον επόμενο γύρο. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες που θα πρέπει να ρυθμιστούν στο θεσμικό ζήτημα αλλά και εδώ ελπίζουμε θα ολοκληρώσουμε το εμπορικό, το εμπορικό πυλώνα επίσης μετά από τόσα χρόνια, 20 χρόνια, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε και την αξιοπιστία μας. Merci, euh, Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στην Μπεατρή Λεγκέικη Καρντόκη, συνέτερο στο Γραφείο Νομικών και Οικονομικών Συμβουλών SAI, πρώην Υφυπουργό Εξωτερικού Εμπορίου στο Υπουργείο Οικονομικών του Μεξικού. Καλησπέρα σα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Μαρία Μερσέντε Ροντρίκερ, καθώ επίση και την Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πρόσκλησή σα αυτή. Ο κόσμος μας γίνεται όλο και πιο πολύπλοκος, όλο και πιο πολυσύνθετος. Δεν, δεν ξέρω αν θυμάστε όταν στα μέσα της δεκαετίας του 90 αρχίσαμε να στέλνουμε τα πρώτα email. Τότε οι επιχειρήσεις αποφάσισαν να κατακαιρματίσουν περισσότερο τις παραγωγικές τους διαδικασίες και να αρχίσουν να παράγουν εκεί πέρα που ήταν πιο φτηνά τελικά για να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και έτσι άλλαξαν και ενδυναμώθηκαν τελικά οι παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Δεδομένων των αλλαγών αυτών που επέφερε αυτή, αυτή η επανάσταση της πληροφορικής, βλέπετε και στη διαφάνεια αυτή ότι το παγκόσμιο εμπόριο άλλαξε δραστικά στον αιώνα μας αυτό από ένα, από ένα εμπόριο προϊόντων σε ένα εμπόριο τελικά που έχει να κάνει με σημαντικές πλέον εισρωές περισσότερο και βλέπετε πως έχουν αυξηθεί όλο και περισσότερο οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών από 42 το 1994 σε 279 το 2018. Δημιουργείται κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν μια πολυπλοκότητα. Διάβασα ένα βιβλίο το οποίο φέρει τον τίτλο Simple Rules, απλοί κανόνες και λένε ότι με ένα τουβλάκι Lego κάνει κανείς ένα συνδυασμό με τρία τουβλάκια 150 1.560 διαφορετικούς συνδυασμούς, ενώ με 6 τουβλάκια λέγκο χάρη στους υπολογιστέ, μπορούμε να έχουμε 900, 915 εκατομμύρια, 915 εκατομμύρια διαφορετικούς συνδυασμούς. Ζούμε λοιπόν σε έναν κόσμο όπου θα μπορούσαμε να πούμε ότι κατά αυτόν τον τρόπο λειτουργούν και συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών και συμβάλλουν σε αυτή την πολυπλοκότητα. Σύμφωνα με το βιβλίο αυτό, Simple Rules, τους απλούς κανόνες, η λύση λοιπόν για έναν πολύπλοκο τέτοιο κόσμο δεν είναι πολύπλοκες λύσεις, αλλά απλοί κανόνες. Και το πιο σημαντικό στο εμπόριο είναι οι κανόνες αυτοί που έχουν να κάνουν με δημόσιες πολιτικές να είναι ουσιαστικά λίγοι, όχι πάνω από πέντε όχι πάνω από πέντε. Πρέπει να ισχύουν πέντε απλοί κανόνες στο παγκόσμιο αυτό εμπόριο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην συγχαίουμε τους απλούς κανόνες με τις απλουστευτικές λύσεις. Πράγμα το οποίο βλέπουμε να ισχύει όλο και περισσότερο τη σήμερον ημέρα με τις λαϊκιστικές κυβερνήσεις. Ένα παράδειγμα είναι ο Ντόναλτ Τραμπ, ο οποίος θεωρεί ότι στρεφόμενος κατά του πολυμερούς εμπορικού συστήματος και κατά των συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου, ξαφνικά θα εξαφανιστούν όλα τα δεινά της αμερικανικής οικονομίας και θα θεραπευτούν όλες οι ασθένειές της. Ας είμαστε λοιπόν πάρα πολύ προσεκτικοί. Και ουσιαστικά ο πρόεδρος Τραμπ αντιμετωπίζει κατά αυτόν τον τρόπο και τη μετανάστευση, θέλοντας να κτίσει απλώς ένα τείχος. Ευτυχώ όμω στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε τον Ντόναλτ Τούσκ, ο οποίο έχει εντελώ διαφορετική προσέγγιση. Απουσία λοιπόν μια ηγετική πλέον από τι Ηνωμένε Πολιτείε είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Λατινική Αμερική να ενισχύσουν ε, τι πολιτικέ και εμπορικέ του σχέσει. Βλέπετε ότι υπάρχουν εδώ πέρα δύο σημαντικοί κανόνες τους οποίους σας προτείνω. Πρώτον, να έχουμε μία όλο και μεγαλύτερη οικονομική ολοκλήρωση. Το Μεξικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό ακριβώς κατάφεραν να πετύχουν πολύ πρόσφατα, όπως ακούσαμε. Και πιο συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό κατάφεραν να, να σημειώσουν πρόοδο στον εξυγχρονισμό τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Μεξικού. Κατάφεραν κατά αυτόν τον τρόπο, αν μου το επιτρέπετε, να βαθύνουν την αγάπη του και να ανανεώσουν του όρκου του. Το προχωρήσουμε σε αυτή τη διαφάνεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίση να σας πω ότι το Μεξικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφεραν να ολοκληρώσουν τον εξυγχρονισμό αυτό πάρα πολύ γρήγορα. Όταν υπάρχει πολιτική βούληση λοιπόν όλα μπορούν να επιταχυνθούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό να αποτελέσει πηγή έμπνευση και για τις υπόλοιπες διαπραγματεύσει στο πλαίσιο της ΝΑΦΤΑ. Έτσι λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό έχουν στείλει ένα πολύ θετικό μήνυμα στον υπόλοιπο κόσμο όσον αφορά την ανοιχτή αυτή στάση στο εμπόριο. Βλέπετε εδώ πέρα τι εμπορικές και επενδυτικέ ροές ανάμεσα στο Μεξικό και την Ευρωπαϊκή Ένωση από τότε που υπεγράφει η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών και τέθησε ισχύ. Το Μεξικό έχει εμπορικό έλλειμμα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά εμείς δεν βλέπουμε τον κόσμο όπω τον βλέπει ο Ντόναλτ Τραμπ. Θεωρούμε ότι οι συναλλαγέ αυτές ήταν πάρα πολύ θετικές από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μας κάναν τελικά πολύ πιο ανταγωνιστικούς σε σχέση με τους υπόλοιπου εταίρου των ΗΠΑ. Ένα 40% των ε, άμεσων ξένων επενδύσεων που φτάνουν στο Μεξικό προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια όμως τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών μειώσαμε τι αρνητικές επιπτώσει τη διάβρωση των προτιμήσεων και δημιουργήσαμε επίση και κάποιου νέου τομεί νέα γενιά στην εμπορική αυτή συμφωνία που αποτελούν βασικά και τι σημαντικότερε προκλήσει στη σύγχρονη οικονομία και επίση καταφέραμε να εμβαθύνουμε τη συμφωνία αυτή σε άλλου τομεί όπω η γεωργία, υπηρεσίε και επενδύσει. Ο πρώτο σημαντικό κανόνα λοιπόν είναι η εμπορική ολοκλήρωση. Ο άλλο σημαντικό όμω κανόνα για να ενισχυθεί η αγάπη μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Μεξικού είναι η σχέση μεταξύ Λατινικής Αμερικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη συνεργασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πραγματικά να υπάρχει μία νομισματική, αν θέλετε, χρηματική αποτίμηση στα όσα λέμε, πραγματικά να επενδύουμε στα όσα διακηρύσουμε ότι θα κάνουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πόσο έχει συμβάλει στην οικονομία της Λατινικής Αμερικής η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως στα πλαίσια των περιφερειακών στρατηγικών και συνεργαζόμενοι με χώρες όπως η Αργεντινή, η Βραζιλία και το Περού. Όσον αφορά τους δύο άλλους τομείς επί των οποίων θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε είναι να αντιμετωπίσουμε τα προστατευτικά μέτρα των ΗΠΑ και από κοινού αυτή τη στιγμή εφαρμόζουμε αντίμετρα κατά των δασμών που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένε Πολιτείε στο αλουμίνιο και τον χάλιβα. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο Καναδά, το Μεξικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση, έχουν τις ίδιες προθέσεις και πραγματικά ελπίζω και οι υπόλοιπε χώρες που έχουν περάσει από διμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με εμά θα ακολουθήσουν αυτή την άγουσα. Κατά αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσουμε ένα πολύ πιο ισχυρό μέτωπο. Επίση θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεργαστεί ακόμα πιο στενά με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής προκειμένου να δημιουργηθεί μια πιο ευρία εμπορική ολοκλήρωση, μια εμπορική συμφωνία πιο ολοκληρωμένη σαν αυτό το οποίο είχε προταθεί πριν από μερικά χρόνια. Πρέπει πραγματικά όμω τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρεθεί πραγματικά σε ηγετική θέση και να, πάρει, να καλύψει αστικά το κενό που έχουν αφήσει οι Ηνωμένε Πολιτείε, οι οποίε στο παρελθόν είχαν προτείνει τη σφαιρική αυτή συμφωνία με τη Λατινική Αμερική. Τέλο, θα ήθελα να αναφερθώ και σε μία μελέτη την οποία εκπώνησε το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ και που είχε να κάνει με την ετοιμότητά μας σε σχέση με το μέλλον της παραγωγής, του παραγωγικού μοντέλου. Και εδώ πέρα πραγματικά πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τις σημαντικότερες προκλήσεις της Επανάστασης 4.0. Στη μελέτη λοιπόν αυτή αντιμετωπίζουμε δύο στοιχεία. Τη διάρθρωση καταρχά της παραγωγής, εδώ αναφερόμαστε περισσότερο στην πολυπλοκότητα και τις δεξιότητες με συγχωρείτε, scale, την κλίμακα. Θέλουμε πραγματικά εδώ πέρα να δούμε πόσο παράγουμε σε, ε, ως προς το ΕΠ και έπειτα η πολυπλοκότητα του νέου παραγωγικού μοντέλου και αυτό μας έχει απασχολήσει. Και μία άλλη συνιστόσα είναι οι κινητήριες δυνάμεις της παραγωγής σε κάθε χώρα, πόσο έτοιμες τελικά είναι οι χώρες. Στις χώρες της Λατινικής Αμερικής βλέπουμε μία δυναμία όσον αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο, την ε, καινοτομία, το θεσμικό πλαίσιο. Θα έλεγα ότι εδώ πέρα πραγματικά μπορούμε να βελτιώσουμε περισσότερο τα πράγματα. Η μελέτη αυτή ταξινομεί τις, τις χώρες αυτές τις εξής κατηγορίες. Τις χώρες οι οποίες βρίσκονται σε ηγετική θέση, οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία. Είστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσετε το μέλλον όσον αφορά τη νέα τεχνολογία. Έχουμε πει τα πιο ιστορικές παλαιότερες οικονομίες και χώρες, όπως το Μεξικό, που υπάρχει μια ισχυρή παραγωγική βάση. Παρόλα αυτά έχουμε χαμηλές επιδόσεις στις βασικές συνιστώσεις της παραγωγής και θα πρέπει να αποφύγουμε να βρεθούμε στριμωγμένοι, αν θέλετε, ανάμεσα στι ε, χώρες που βρίσκονται στη ηγετική θέση και τι αναδυόμενε χώρες που προτείνουν χαμηλότερο εργατικό κόστο. Οι άλλε δύο κατηγορίε είναι οι χώρε με υψηλό δυναμικό, οι οποίες έχουν περιορισμένη παραγωγική βάση, αλλά έχουν ένα πολύ καλό δυναμικό όσον αφορά τις κινητήρες παραγωγικές δυνάμεις και έπειτα έχουμε και τις αναδυόμενες χώρες, τις εκολαπτώμενες αγορές, όπου εκεί έχουμε και τις περισσότερες χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπου έχουμε περιορισμένη παραγωγική βάση και χαμηλέ επιδόσει όσον αφορά τι βασικέ συνιστώσει παραγωγή. Κατά αυτόν τον τρόπο ταξινομούνται οι χώρε σε αυτή τη μελέτη και με μπλε εδώ πέρα βλέπετε τι χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση που βρίσκονται σε ηγετική θέση και με κίτρινο βλέπετε τις χώρες της Λατινικής Αμερικής οι οποίες βρίσκονται ουσιαστικά στην κατηγορία των αναδυόμενων οικονομιών. Μόνο το Μεξικό βρίσκεται στην κατηγορία legacy countries, πιο παραδοσιακές αν θέλετε οικονομίες. Τέλος, όσον αφορά το τι θα πρέπει να κάνει το Μεξικό και εν γέννη Λατινική Αμερική και εν γέννη τι πρέπει να κάνουμε και σε παγκόσμιο επίπεδο. Θέλουμε να υιοθετήσουμε το πλέον κατάλληλο οικονομικό μοντέλο και την κατάλληλη οικονομική εμπορική πολιτική. Θα πρέπει να μα απασχολήσει προφανώ το ζήτημα τη παραγωγικότητα, προκειμένου να επιλύσουμε προβλήματα ανισοτήτων, τα οποία τα βλέπουμε όλο και περισσότερο στι οικονομίε μα. Στην περίπτωση του Μεξικού, όπω βλέπετε και στη διαφάνεια, έχουμε καταφέρει να μειώσουμε, έχουμε μια μείωση μάλλον στην παραγωγικότητα και αυτό αντικατοπτρίζεται στο κατακεφαλή ΝΑΕΠ σε σχέση με χώρες όπως η Κίνα για παράδειγμα, όπου εκεί έχουμε αύξηση. Ακολουθώντας λοιπόν τους απλούς κανόνες που σας περιέγραψα στην αρχή της παρουσίασής μου, αυτοί θεωρώ ότι είναι οι πέντε απλοί κανόνες οι οποίοι θα αλλάξουν πραγματικά τα πράγματα προς το καλύτερο στη Λατινική Αμερική. Να έχουμε έναν καλύτερο παραγωγικό μετασχηματισμό, προκειμένου να προσανατολιστούμε προ δραστηριότητε υψηλότερη αξια Το προσωπάκι αυτό που χαμογελάει, βλέπετε εδώ πέρα όλη την αλυσίδα παραγωγη η οποία δημιουργεί αυτή την καμπύλη του χαμογέλου εδώ. Όσο πιο κοντά φτάνει κανεί στι γωνίε, τόσο μεγαλύτερα είναι και προστιθέμενη αξία. Δυστυχώ το Μεξικό βρίσκεται αρκετά χαμηλά στο μεταποιητικό τομέα. Θα πρέπει να καταφέρουμε εκεί πέρα να επενδύσουμε περισσότερο να επενδύσουμε περισσότερο στην έρευνα και την καινοτομία, να ασχοληθούμε με τη χρήση εμπορικών σημάτων και έπειτα υπάρχουν και άλλε συνιστώσει όπω το μάρκετινγκ, η διανομή και οι πωλήσει. Και βλέπετε εδώ πέρα πώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βοηθήσει το Μεξικό να καταφέρουμε να διασυνδέσουμε μικρομεσαίες επιχειρήσει με πολυεθνικέ επιχειρήσει για να συμμετέχουμε περισσότερο σε παγκόσμιε και περιφερειακέ αλυσίδε αξιών, σε δεύτερο λόγο θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην καινοτομία και να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες δεξιότητες για τις ανάγκες της αγοράς. Θα πρέπει να καταφέρουμε να αυξήσουμε το παραγωγικό μας μοντέλο, να λειτουργούμε πιο γρήγορα και με χαμηλότερο κόστος και θα πρέπει να βελτιώσουμε επίσης και την, το συντονισμό ανάμεσα στον ιδιωτικό, το δημόσιο φορέα και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και ξέρω ότι ως προς αυτό έχει βοηθήσει ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση της κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής, να γίνει δηλαδή αυτή η διασύνδεση ανάμεσα σε επιχειρήσεις και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Είμαι πεπισμένη ότι μέσω της συνεργασίας και μέσω των στρατηγικών διαπραγματεύσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη, με τη βοήθειά σας λοιπόν θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε περισσότερο σε ένα μοντέλο το οποίο θα αυξήσει τον παραγωγικό και μεταποιητικό κλάδο στη Λατινική Αμερική. Μαρία Γκαρθία από το Πανεπιστήμιο του Μπαθ. Ε, μέσω τηλεδιάσκεψης. Okay. Uh, good afternoon. Uh, can you hear me okay?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 από την Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου του Μονάχου. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Μου ζητήθηκε να μιλήσω για το Μερκοσούρ και τη νέα πνοή και τις δυνατότητες αυτής της συμφωνίας. Λοιπόν, τέσσερις χώρες, Αργεντίνη, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουάη είναι 150 εκατομμύρια εργαζόμενοι, 250 εκατομμύρια καταναλωτές. Είναι η μεγαλύτερη, η μεγαλύτερη περιοχή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ελευθερού εμπορίου. Ε, βέβαια τον κύριο ρόλο τον παίζει η Βραζιλία, οι άλλες χώρες ε, είναι μικρότερες η περιοχή έχει θέματα πολιτικής σταθερότητα και μακροοικονομικής σταθερότητα, οπότε η επιτυχή κατάρριξη της Συμφωνίας ε, Ένωση ε, Μερκοσούρ θα μπορούσε να βοηθήσει τη σταθερότητα ε, της περιοχής και να αναχαιτήσει τον οικονομικό λαϊκισμό. Μερικά στοιχεία οικονομικά. Η Βραζιλία μόλις βγαίνει από την βαθύτερη ύφεση της ιστορίας της. μειώθηκε κατά 7% περίπου το ΑΕΠ μεταξύ 15 και 17. Η Αργεντινή διέρχεται κρίση. Μόλις ε, δέχθηκε ένα πρόγραμμα του ΔΝΤΑΦ έχει πληθωρισμό 85%. Άρα είναι σε περιδίνηση, μακροοικονομική περιδίνηση. Η διατάραξη. Η Παραγουάη ακόμη θεωρείται αναπτυσσόμενη χώρα. Έχει λοιπόν ακόμη, υπάρχει ακόμη στο GSP sin της Ένωσης. Μια ερώτηση που θέτουν οι οικονομολόγοι όταν εξετάζουν εμπορικέ συμφωνίες είναι τι δυνατότητες έχει μια συμφωνία ελευθέρων των Πόσο θα, πόσο θα αυξηθούν οι εξαγωγές και άρα πόσο θα εκτονώσει την οικονομία. Για παράδειγμα, για να δούμε πόσο είναι οι εξαγωγές σε σχέση με το ΑΕΠ. Αργεντινή και Βραζιλία περίπου το ίδιο. Αλλά αν συγκρίνουμε με χώρες που είναι στο ίδιο επίπεδο ανάπτυξης, περίπου το ίδιο μέγεθος, μιλάει την ίδια γλώσσα και έχει εμπορική συμφωνία με το, την Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπετε πόσο μεγάλη είναι η διαφορά. Το Μεξικό είναι σχεδόν 40% οι εξαγωγέ του ΑΕΠ. Άρα υπάρχει πολύ περιθώριο για περαιτέρω εμπόριο. Και αν ε, συγκρίνουμε με μια παρόμοια χώρα, από πλευρά μεγέθου και επίπεδο ανάπτυξη, την Τουρκία, βλέπουμε λοιπόν ότι η Αργεντινή και η Βραζιλία υπολείπονται. Τώρα μπορούμε να κάνουμε περαιτέρω στατιστική ανάλυση. Αλλά τουλάχιστον ε, μπορούμε να εξαγάγουμε το συμπέρασμα ότι υπάρχει πολύ αναξιοποίητο δυναμικό μεταξύ Ευρώπης και Μερκοσούρ. Πρόσφατες ε, τώρα στατιστικές συναλλαγών. Ένωσης Μερκοσούρ. Βλέπουμε διακυμάνσεις. Η μπλε γραμμή πάνω-πάνω είναι οι εξαγωγές της Ένωσης προς την περιοχή Μερκοσούρ. Και η βάση είναι 100 το 2002. Έχει υπάρξει μεγάλη ανάπτυξή τους. Έχουν ε, πολλαπλασιαστεί επί 2,5. Θετικό αυτό. Τώρα όμως οι εξαγωγές του Μερκοσούρ. Οι εισαγωγές στην Ένωση δεν είναι τόσο εντυπωσιακή ανάπτυξη. Εμείς εξάγουμε 44 δις, εισαγωγές 42 δισεκατομμύρια, αλλά ένα μικρό πλεόνασμα για την Ένωση. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε περιόδους ε, εκρηκτικής ανάπτυξης ε, και έντονης κρίσης. Έχει να κάνει με τις τιμές των πρώτων υλών που ε, διακυμαίνονται πολύ οι συμφωνίε Ένωση Μερκοσούρ θα μπορούσαν να βοηθήσουν την περιοχή να εξάγει και άλλα προϊόντα για να υπάρξει σταθεροποίηση του μακροοικονομικού κύκλου. Και τώρα ποσοστό αγοράς στο Ινστιτούτο μας, IFO, ιδιαίτερα στην περιοχή Μερκοσούρ, η Κίνα εξάγει όλο και περισσότερο και κατά πάσα πιθανότητα ή το 17 ή το η Κίνα θα μετατραπεί στον πρώτο εμπορικό εταίρο της περιοχής, άρα και περισσότερο πολιτικό βάρος. Οπότε μια συμφωνία δική μας με τον Μερκοσούρ θα μπορούσε να αναστρέψει αυτή την πορεία. Η περιοχή αυτή έχει πολύ υψηλές, πολύ υψηλούς παγιοποιημένους δασμούς. Είναι διψήφιοι μπορεί να πάνε μέχρι 35%. Τα αυτοκίνητα για παράδειγμα που εξάγονται από την Ευρώπη στη Βραζιλία υφίστανται δασμό 35. Από την άλλη μεριά οι εφαρμοζόμενοι δασμοί είναι χαμηλότεροι. Βλέπετε εδώ ότι είναι λιγότερο κόκκινα τα χρώματα. Δεν είναι τόσο υψηλή αυτή η δασμή. Τι σημαίνει αυτή, είναι ότι σηκώνει νερό το φαινόμενο. Ξέρετε ότι οι παγιοποιημένοι δασμοί είναι αυτοί που εγγυώνται οι συμφωνίες ε, του ΠΟΕ, ενώ οι εφαρμοζόμενοι είναι αυτοί που εφαρμόζονται. Αυτό έχει κάποιες επιπτώσεις. Ναι, μεν υπάρχουν ε, υψηλοί δασμοί, ενώ οι δικοί μας ε, εισαγωγικοί δασμοί είναι πολύ χαμηλότεροι. Άρα εκείνοι πρέπει να μειώσουν τους δασμούς τους. Άρα θα ωφεληθούμε. Πρέπει να ανοίξει πολύ περισσότερο τις αγορές του το Μερκοσούρ από ότι η Ευρώπη. Και οι πολυμερείς ε, ταρίφες του Μερκοσούρ είναι υψηλές. Άρα, εάν βάλουμε το πόδι στην πόρτα της περιοχής, τότε θα ωφεληθούν πολύ οι δικοί μας παραγωγοί. Η παραγωγή της Κίνας ή των ΗΠΑ δεν θα έχουν τέτοια προνομιακή μεταχείριση. Άρα αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ σκόπιμο κάτι τέτοιο για μας. Άρα θα ωφεληθούμε από αυτόν που πρωτομπαίνει σε μια αγορά. Και τα αποτελέσματα απόκ... Ε, απόκλησης του εμπορίου, ε, μάλλον διαφοροποίησης του εμπορίου θα μπορούσε να μας βοηθήσει περισσότερο το γεγονό ότι οι παγιοποιημένοι από του εφαρμοζόμενου, από δασμού είναι τόσο διαφορετικοί σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα. Εκτό τη Αφρική, αυτή είναι η περιοχή όπου υπάρχουν περισσότερε αβεβαιότητε για του Ευρωπαίου εξαγωγεί. Οι χώρε Μερκοσούρ μπορούν να αλλάξουν ε, του δασμού του ε, στον ΠΟΕ όποτε θέλουν. Και για κάποια περίοδο, 400 περίπου από τις 5.000, ε, θα μπορούσαν και να τριπλασιάσουν τους δασμούς τους αν θέλουν. Μια συμφωνία θα ε, καταργούσε αυτή την αβεβαιότητα. Άρα αυτό θα μας δημιουργήσει περισσότερες δυνατότητες εξαγωγών γιατί εδώ υπάρχει τόση αβεβαιότητα. Και η Ευρώπη έχει λεπτά θέματα ιδιαίτερα στον τομέα του βοήου, της ζάχαρης, των ε, σπορελαίων, της βιοεθανόλης. Οπότε και οι δύο πλευρές θα χρειαστούν μεταβατικές περιόδους και ποσοστώσεις για τα πιο ευαίσθητα προϊόντα τους. Τώρα η μη δασμολογική φραγμή. Πολλά θέματα έχουν σημειώσει διάφορες μελέτες. Η Παγκόσμια Τράπεζα μας λέει ότι και οι τέσσερις αυτές χώρες δεν τα πάνε πολύ καλά όσον αφορά τις τελωνιακές διαδικασίες, πολύ γραφειοκρατικές και χρονοβόρες και ενέχουν κινδύνους για τους εξαγωγείς μας. Άρα αν βελτιωθεί η κατάσταση θα βοηθήσουμε πολύ τους εξαγωγείς μας. Επίσης ε, διακρίσεις για τους φόρους. Εισαγωγές ε, περιορισμένες, περιορισμένες εισαγωγές στην Αργεντινή. 26% των προϊόντων που εισάγει η Αργεντινή θεωρούνται ευαίσθητα και χρειάζονται ειδικέ άδειε. Για παράδειγμα, χρειάζεται διπλή πιστοποίηση σε κάποιους κλάδους. Έχουμε προβλήματα με τις ε, υγειονομικές και φυτο ε, προδιαγραφές, ιδιαίτερα για το κρέας και το ψάρι. Και για τις δημόσιες προμήθειες υπάρχει νομοθεσία που ευνοεί τους ε, τοπικούς συμμετέχοντες. Επίσης ε, η προστασία των ε, πνευματικών δικαιωμάτων. Η Βραζιλία δεν έχει υπογράψει ε, κάποιες συμφωνίες και υπάρχουν και κάποιες, κάποιοι φραγμοί για τις επενδύσεις. Προσπαθήσαμε να βάλουμε αριθμούς, να κάνουμε εκτιμήσεις για τι σημαίνουν η άρση, τι θα σήμαινε η άρση αυτών των περιορισμών. Θεωρούσαμε ότι αν υπάρχει κάτι τέτοιο θα μπορούσαμε να αυξήσουμε το ΑΕΠ μας μεταξύ 0,07 και 0,18 σε δισεκατομμύρια είναι 10 έως 25 δις επιπλέον ΑΕΠ στην Ευρώπη. Για τις χώρες του Μερκοσούρ θα σήμαινε κάτι παρόμοιο είναι 12 με 34 ευρώ επιπλέον αλλά το ποσοστό που διαπιστώνεται εδώ είναι πολύ ψηλότερο από το ευρωπαϊκό. Οι χώρες αυτές θα το ιδιαίτερα. Βέβαια θα μειωθεί το δασμολογικό εισόδημά μας περίπου ένα δις. Θα είναι πολύ διαφορετική κατάσταση από χώρα σε χώρα. Για τις χώρες του Μερκοσούρ θεωρούμε ότι η Παραγουάη και η Ουρουγουάη... θα ωφεληθούν περισσότερο από την Αργεντινή και την Βραζιλία γιατί είναι μικρότερες και εξαρτώνται περισσότερο από το διεθνές εμπόριο. Και στην Ευρώπη θα είναι μεγάλη ανισορροπία. Οι ισπανικές χώρες της Ένωσης η Ισπανία και η Πορτογαλία θα ωφεληθούν περισσότερο από τις χώρες του κέντρου της Ευρώπης. Τώρα, ανακλάδο. Τι επιπτώσει θα έχει μια τέτοια συμφωνία. Είναι κλασική περίπτωση χωρών που ε, ειδικεύονται σε διαφορετικούς τομείς. Εμείς έχουμε πλεονέκτημα στην, ε, στον κατασκευαστικό κλάδο, και είναι στον γεωργικό. Άρα είμαστε συμπληρωματικοί. Οι περισσότεροι κατασκευαστικοί κλάδοι θα ωφεληθούν, θεωρούμε, και τα δίκτυα θέμες αξίας εντός της ε, ενιαίας αγοράς θα έχουν ως επίπτωση ότι η αύξηση των εξαγωγών της Γερμανίας για παράδειγμα θα επιφέρει ωφέλη και σε άλλες χώρες για παράδειγμα στην κεντρική Ευρώπη κυρίως. Κάποια άλλη κλάδη είναι πιο ε, ευάλυτη. Έχουμε εδώ την ξυλία, τα έπιπλα, το χαρτί, τα κλωστοφαντουργικά και το δέρμα. Αλλά θα κερδίσουμε πολλά σε βασικούς γεωργικούς ε, υποκλάδους. Είπαμε κρέας, ε, ζάχαρη, σπορέλαια, βιοεθανόλια. Αλλά όλα θα εξαρτηθούν από τις λεπτομέρειες μετά τις ε, συμφωνίες, τις οποίες φυσικά δεν έχουμε. Επίσης υπάρχουν ευκαιρίες ιδιαίτερα και στον γεωργικό τροφιμικό τομέα, το γάλα και άλλο όπως είναι για παράδειγμα ο λυκίσκος και τα σπαράγγια. Πολλές μελέτες έχουν βεβαιώσει ότι θα ωφεληθούν όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης και η προστιθέμενη αξία στο κατασκευαστικό κλάδο αντισταθμίζει και υπερσκελίζει κατά πολύ τις ε, απώλειες στον ε, γεωργικό τομέα. Και μάλιστα μπορεί και να υποτιμούμε το πραγματικό αποτέλεσμα της αύξησης των ε, εμπορικών ροών γιατί είναι πολύ ψηλές, ε, πολύ υψηλοί δασμοί και θα καταργούσαμε την αβεβαιότητα. Είναι δύσκολο τώρα να κάνεις μια ε, αριθμητική εκτίμηση των αποτελεσμάτων και αναμένουμε και θετικά αποτελέσματα για την μακροοικονομική σταθερότητα της περιοχής αυτής. Αυτό θα ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις, αλλά δύσκολο να προβλέψουμε σε τι βαθμό. Και επίσης ε, υπάρχει ε, και ουσιώδης αβεβαιότητα όσον αφορά το, τη μείωση του κόστους του εμπορίου λόγω της μείωσης των δασμών. Και ορισμένα άλλα συμπληρωματικά αναμένουμε ότι η συμφωνία αυτή θα δημιουργήσει προβλήματα για κάποιους ε, τομείς στον τομέα το γεωργικό και των τροφίμων στην Ευρώπη Πρέπει να το λάβουμε υπόψη όταν θα αναθεωρήσουμε την κοινή γεωρική πολιτική και όταν θα ζητήσουμε το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Ίσως θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε πόρους από το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για να βοηθήσουμε τη γεωργία μας. Υπάρχουν ανησυχίε για τις επιπτώσεις των συμφωνιών για τα αέρια θερμοκηπίου και τη βιοπικιλότητα. Είναι όντως ε, εξωτερικές επιπτώσεις αυτές, εξωγενείς. Πρέπει λοιπόν η συμφωνία αυτή να μην συμβάλλει στην περαιτέρω αποψήλωση στη Βραζιλία και την Παραγουάη. Πρέπει να υπάρχει επιτήρηση πραγματικό χρόνου για να μην έχουμε παράπλευρες απώλειες που είναι απόλυτα ανεπιθύμητες. Αλλά πρέπει η πολιτική που θα ακολουθήσουμε για τα βιοκάψιμα στην Ευρώπη να μην προκαλέσει διακρίσεις. Υπάρχουν τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των μειονοτήτων και των γηγενών πληθυσμών. Και όλα αυτά μας ανησυχούν ουσιοδό. Αν και είναι πολύ μακριά από αυτά που πρέπει να σας εξηγούν οι οικονομολόγοι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Προτείνω να περάσουμε στις ανταλλαγές ε, απόψεων με τα μέλη μας. Θα δώσω το λόγο στον μόνιμο εισηγητή για την Λατινική Αμερική καταρχήν, τον κύριο Φίσας, που είναι υπεύθυνος για την Κολομβία και το Περού. Ε, muy bien, eh, Βρισκόμαστε στο στάδιο της εφαρμογής ε, της Εμπορικής Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κολομβία και Περού. Αυτό δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή ή είναι αργότερα αυτό. Sí, no, no es ahora. Όχι τώρα, ε. Καλά το κατάλαβα. Je vais donner... Θα δώσω το... Θες να πεις κάτι τώρα? Οκ. Okay. Ο λόγος στην κυρία Δοντρέγκο Πινιέρο. Χαίρομαι που λαμβάνει η χώρα αυτή η ακρόαση. Είναι μεγάλη ευκαιρία για να υπογραμμίσουμε την ε, σημασία που αποδίδει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γενικότερα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις σχέσεις πολιτικές, οικονομικές και εμπορικές με την Λατινική Αμερική. Θέλω να υπογραμμίσω ότι πέραν των ιστορικών και πολιτιστικών δεσμών που μας ενώνουν και πέραν των αρχών και των αξιών που μοιραζόμαστε, συνεργαζόμαστε πολύ στενά σε πολλά πολυμερή φόρα, ακριβώς για να προσπίσουμε αυτές τις αρχές υπέρ ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ε, περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, ε, πολύ πιο σημαντικά από ό,τι παλιότερα. Γιορτάζουμε σήμερα την Παγκόσμια ημέρα των προσφύγων και γνωρίζουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ εγκατέλειψε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Όμως εμείς με τη Λατινική Αμερική συνεργαζόμαστε ε, προσπίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό είναι που πρέπει να προϋπογραμμίσουμε πάνω από όλα και πάνω από τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις, όσο σημαντικές και αν είναι αυτές. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις, θέλω να σημειώσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Λατινική Αμερική μαζί αντιπροσωπεύουμε το 25% του παγκοσμίου ΑΕΠ και το 25% του παγκόσμιου πληθυσμού. Οπότε στην ε, πολιτική και την οικονομική ατζέντα η Λατινική Αμερική παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο ε, στις διαπραγματεύσεις και αυτό είναι πολύ θετικό. Σε ό,τι αφορά την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό, ακούσαμε τις παρουσιάσεις ε, πολύ πλήρεις ε, και από τις δύο κυρίες. Ε, θέλω όμως να εφιστήσω την προσοχή σας στο εξής. Πρόσφατα ήμασταν σε αποστολή στο Μεξικό και έχω την εντύπωση ότι ήταν πολύ κρίσιμη κέρια αυτή η επίσκεψη γιατί το Μεξικό βρίσκεται το μέσο μιας προεκλογικής διαδικασίας και θέλαμε να μάθουμε ποια είναι η άποψή τους, η άποψη των υποψηφίων αλλά και ποια είναι και η άποψη της κοινωνίας σε σχέση με τη συμφωνία αυτή και μπορώ να σας ενημερώσω ότι επικρατεί μια ομοφωνία μεταξύ των πολιτικών ομάδων σε ό,τι αφορά την στήριξη τη συμφωνίας. Προφανώς υπάρχουν κάποια θέματα που είναι κρεμή ακόμα. Θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες από όλους από πλευρά του Μεξικού για να ρυθμιστούν και αυτά. Για παράδειγμα, κρατικές, ε, άνοιγμα των κρατικών ε, ε προμηθειών σε επίπεδο ε, περιφερειακό πριν τελειώσει το έτος Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να επικυρωθεί το, η Σύμβαση 98 ε, του Παγκοσμίου Οργανισμού Εργασίας. Ο κ. Φίσας εκ μέρους του ΕΛΚ και εγώ ίδια ε, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον Υπουργό Εργασίας ε, ο οποίος μας ανέφερε ότι το Μεξικό ε, έχει αποφασίσει ήδη την παραπομπή του θέματος της ε, Σύμβασης 98 στη Γεωσία, όπου και θα επικυρωθεί. Ε, και τους είπαμε ότι καλό είναι αυτό που γίνεται, διότι θα είναι προς του Μεξικού. Σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υπάρχει ένα ειδικό κεφάλαιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και είναι μάλιστα και το πρώτο με αυτή την ιδιαιτερότητα. Πρέπει να κάνουμε αυτή την προσπάθεια και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό έτσι ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να είναι ενήμερες όλων των πλέον προκύπτουν από τη συμφωνία. Χρειάζεται όμως να το προσπαθήσουμε. Όλες οι επαφές ε, τις οποίες είχαμε με τους υπεύθυνους επιχειρηματίες κλπ. μας ε, ε, έπεισαν ότι αυτό πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να προβάλλουμε τα κέρδη και τα ωφέλη που προκύπτουν. Οι προτιμήσεις χρησιμοποιούνται σε πολύ μικρό ποσοστό. Δεν έχει κανένα νόημα να υπογράφουμε μια συμφωνία και τελικά ε, οι προτιμήσεις οι οποίες προβλέπονται ε, να τη χάνουν χρήσεις μόνο κατά 50%. Δεν έχει κανένα νόημα. Πρέπει να φτάνουμε το 100%. Μετά την σύναψη λοιπόν της συμφωνίας θα πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε να εφαρμοστεί κάθε ολοκληρία. Μόνο έτσι θα πετύχουμε τους στόχους μας. Σε ό,τι αφορά το θέμα του φύλου, είναι αλήθεια ότι η εντολή για τις διαπραγματεύσεις με το Μεξικό δεν περιλάμβανε κεφάλαιο για το φύλλο. Ε, η συμφωνία με τη Χιλή θα είναι η πρώτη που θα περιλαμβάνει τέτοιο κεφάλαιο. Όμως παρόλα αυτά μπορούν να γίνουν πράγματα και να συμπεριληφθούν στη συμφωνία. Χαιρόμαστε που υπάρχει ένα ειδικό κεφάλαιο για την ευημερία των ζώων. Κρίμα που δεν υπάρχει ένα ειδικό κεφάλαιο για το 50% του πληθυσμού που είναι γυναίκες στο πλαίσιο της συμφωνίας, χωρίς να ξανανοίξουμε τα διάφορα κεφάλαια, θέλουμε να εντάξουμε το αποτέλεσμα των μελετών που δείχνουν πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις γυναίκες στη ζωή τους μέσω αυτής της συμφωνίας. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσω για το Μερκοσούρ. Ο κ. Σαλαφράγκα είναι παρόν νομίζω που είναι πιο ειδικό για το θέμα αυτό. Αλλά να πω και εγώ δύο λόγια. Και αυτή η συμφωνία είναι μεγάλη ευκαιρία για μας. Η εντολή χρονολογείται από το 1998 δυστυχώς είναι πάρα πολύ παλιά, απαρχαιωμένη. Έχουμε καινούργιες ε, φιλοδοξίες με τις νέες επικαιροποιημένες συμφωνίες, όμως ε, πρέπει να προχωρήσουμε. Ε, αυτό που με προβληματίζει είναι το εξή. Σε αυτές τις συμφωνίες των οποίων η διαπραγμάτευση θα είναι πολύ περίπλοκη, έτσι παίρνει μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε όλες αυτές τις συμφωνίες θα έπρεπε να έχουμε πιο ευέλικτους μηχανισμούς ε, προκειμένου στο μέλλον να μπορούμε να εντάξουμε καινούριε πτυχές της εμπορικής πολιτικής. Δεν έχει νόημα ε, στο συμφωνία με το Μερκοσού να μην μπορούμε να προβλέψουμε οτιδήποτε ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν συμφωνούμε και οι δύο, γιατί να μην προβλεφθεί για παράδειγμα μια ενιαία θηρίδα και για τις τέσσερις χώρες του Μερκοσούρ και για την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν μπορούμε να προσθέσουμε κάτι για, που να έχει σχέση για παράδειγμα με αυτά που υπογράφηκαν στην Υπουργική ε, Συνάντηση ε, του Buenos Aires για το φύλλο. Αυτό, αυτά, αυτά τα αποτελεσμάτα τα υπέγραψαν οι, χώρε χώρες του Μαρκοσούρ. Είναι αν, ανηληφθήσεις υποχρεώσεις. Γιατί να μην μπορούμε να τα προσθέσουμε αυτά οι πολίτες μας και οι επιχειρήσεις το περιμένουν από μας Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπέγκεν ενδεχομένω θέλει να πάρει το λόγο. Όχι. Εσείς παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις ε, ενδιαφέρουσες ε, παρουσιάσεις. Νομίζω ότι έχουμε εδώ και πολύ καιρό λάβει την εντολή και έχουμε χάσει αρκετό χρόνο. Και θα ήθελα να μάθω πώς εκτιμάτε τη συμβολή του ψηφιακού κλάδου. Επισκεφθήκαμε την Κολομβία και διαπιστώσαμε ότι είναι ακόμη εν τη γενέση, αλλά αρχίζει να αναπτύσσεται ο κλάδος αυτός έστω και με αβέβαια βήματα. Πρέπει λοιπόν, ε, εφόσον ε, θέλουμε οι διαπραγματεύσεις να ανταποκρίνονται στη σημερινή κατάσταση, να συμπεριλάβουμε και αυτό το τομέα και ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες και τις startup. Και όταν έχουμε συνεργασίες, να τίθενται τα θέματα προστασίας δεδομένων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ εσείς. Και εγώ ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις. Ξέρετε όλοι ότι σε μια συμφωνία πάντα υπάρχουν χαμένοι και κερδισμένοι. Βεβαίως στον οικονομικό κλάδο κερδίζουν πολλοί. Ποιοι είναι όμως αυτοί που χάνουν, όπως υπόθηκε και στις παρουσιάσεις. Τι συμβαίνει για παράδειγμα εάν υπογράψουμε τέτοια συμφωνία, τι θα γίνει στην Ήπεθρο, τι θα γίνει με τους αγρότες, τους οποίους τους διώχνουν από τη γη τους, χωρίς καμία προστασία των δικαιωμάτων τους. Και γενικά η κοινωνία των πολιτών δεν εμπλέκεται στη διαδικασία. Συναντηθήκαμε στον Παναμά στα πλαίσια του ε, Ευρωλάτ και συζητήσαμε για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε να συμπεριληφθούν μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλες οργανώσεις αλλά μας υπόθηκε ότι για αυτή την συμφωνία θα μπορούσε να είναι καλύτερη η συμμετοχή τους. Πώς μπορούμε λοιπόν να βελτιώσουμε. Και θέλω να τονίσω ακόμη περισσότερο την βιωσιμότητα. Έχουμε προβλήματα και για τα δικαιώματα των εργαζομένων και για την προστασία του περιβάλλοντος. Πρέπει να υπάρχει ένα ιδιαίτερα ρωμαλαίο και εφαρμόσιμο κεφάλαιο για την ε, βιωσιμότητα. Και να προβλέπει και κυρώσει. Εάν γίνονται παραβιάσει, να υπάρχουν και κυρώσει. Για να το αντιμετωπίσουν σοβαρά οι πάντε. Δεν είναι δυνατόν όλα αυτά θελούσια. Δεν είναι δυνατόν απλώ να γίνονται διακηρύξει και να αναλαμβάνονται δεσμεύσει μόνο στα λόγια. Οι διαπραγματεύσει ε, κρατάνε εδώ και 18 χρόνια. Θέλουμε βεβαίω μια δίκαιη συμφωνία και με τη Μερκοσούρ και με άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Πρέπει λοιπόν και οι δύο πλευρές να είναι αξιόπιστες. Και η Ευρώπη και η Λατινική Αμερική πρέπει να τηρούν τους κανόνες, να συμμετέχει στη διαμόρφωση και τέλος των προγραμμάτων η κοινωνία των πολιτών. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Έχετε ιδέες εσείς ως ομιλητές πώς μπορούμε να βελτιώσουμε περαιτέρω αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Οι συμμετέχοντες στο πάνελ θέλουν να πάρουν ενδεχομένως ε, το λόγο ή κάποιοι άλλοι συμμετέχοντες, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Όντως, η εντολή για τις διαπραγματεύσεις με το Μερκοσούρ ε, είναι 20 ετών. Δεν είναι δυνατόν να διαπραγματευόμεθα με εντολή 20 ετία. Έχει αλλάξει άρδινο κόσμος σε αυτό το διάστημα, άρα είναι απόλυτα αναγκαίο. Αυτά που λέει για παράδειγμα το κείμενο για το εμπόριο για όλους να ληφθούν υπόψη γιατί είναι τόσο παλιά η εντολή. Γι' αυτό θα κάνω μια πρόταση που θα λέει ότι επειδή είναι αυτή η κατάσταση θα διαπραγματευτούμε με βάση αυτή την εντολή αλλά θα υπάρχει 100 προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να εξεχρονιστεί η συμφωνία με βάση μια νέα εντολή για παράδειγμα μέσα σε μια δεκαετία ούτως ώστε θα καταλήξουμε σε μια νέα συμφωνία. Τα συζητήσαμε για τη Χιλή, για το Μεξικό, με τι οποίε χώρε έχουμε συμφωνίε ελευθέρων συναλλαγών, οι οποίε ισχύουν εδώ και αρκετό διάστημα και μα δόθηκε εντολή να υπάρξει τώρα εξυγχρονισμό. Έχουμε λοιπόν μια δυναμική που μας επιτρέπει να καταλήξουμε σύντομα με το Μερκοσούρ για να καλύψουμε μετά και τα άλλα κεφάλαια, ιδιαίτερα στον ψηφιακό τομέα. Μα ενδιαφέρει ιδιαίτερα εμάς εδώ ω Ευρώπη να υπάρξουν ε, κανόνε που να είναι συμβατοί με τους κανόνες μας για την προστασία των δεδομένων με τον νέο βασικό κανονισμό. Έχει αλλάξει τη, τους όρους του παιχνιδιού. Άρα πρέπει και σε αυτές τι διαπραγματεύσεις να ληφθεί υπόψη. Γιατί υπάρχει κίνδυνος ψηφιακού προστατευτισμού δεν είναι θεωρητικός. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο. Αυτό ισχύει και για άλλα σύγχρονα θέματα. Βιωσιμότητα, οπωσδήποτε. Το θέμα της αποψήλωσης, ε, εκπομπές διοξιδίου του άνθρακου, αλλαγή της χρήσης γης. Όλα αυτά είναι βασικά θέματα. Και ακριβώς η συμφωνία με το Μερκοσούρ πρέπει να τα αντιμετωπίσει έστω και αν δεν τα λύσει πλήρω, να δώσει μια προοπτική, ίσω σε ένα δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων να επιληθούν. Δηλαδή, μέσω πρόθεσμα έχουμε και να συζητήσουμε για τέτοιε συμφωνίε με την Ινδονησία. Και εκεί τίθενται ακριβώ τα ίδια θέματα που αφορούν τη Βραζιλία και την Παραγουάη. ψηλό των δασών και αλλαγή τη χρήση γης. Νομίζω ότι πολλοί οικονομολόγοι που ασχολούνται με τα θέματα αυτά θα σας πούν ότι οπωσδήποτε πρέπει να προβλέπει κυρώσεις και το κεφάλαιο βιωσιμότητας. Γιατί το θέμα είναι παγκόσμιο. Ιδιαίτερα όσον αφορά το διοξίδιο του άνθρακος. Άρα χρειαζόμαστε ρωμαλαία κείμενα. Εάν δεν υπάρχουν ε, παγκόσμιες ε, εξωγενείς επιπτώσεις, δεν είναι τόσο προφανές ότι πρέπει να είναι τόσο κατηγορηματικά τα κείμενα, αλλά για το διοξείδιο του, άνθρακο, σίγουρα, άνθρακος σίγουρα πρέπει να συμπεριληφθούν και κυρώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Να μιλήσω κι εγώ στα Ισπανικά, μια και κάποια από, τους, από τα μέλη σας μίλησαν στα Ισπανικά. Το είπα και στην παρουσίασή μου, αλλά ε, ίσως πρέπει να το επαναλάβω. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή της παγκόσμιας οικονομίας. Πρέπει να κερδίσουμε τη μάχη του ελεύθερου εμπορίου. Τη μάχη του μοντέλου που δημιουργήσαμε, που πιστέψαμε και πιστεύουμε θα μας δώσει σταθερότητα, ειρήνη και οικονομική ανάπτυξη για το μέλλον. Παρ' όλα αυτά, στην ανάλυση της παγκόσμιας οικονομίας θα πρέπει να συνεκτιμήσουμε το ότι το γεγονός της οικονομίας αγοράς όπου θεωρούσαμε κάποτε ότι οι αγορές θα λύσουν όλα τα προβλήματα δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει να εμπνεύσουμε στις χώρες μας μια νέα βιομηχανική πολιτική, ε, μια νέα πολιτική ε, ε, δημιουργική παραγωγική πολιτική. Και ο τρόπος ε, είναι να διευρύνουμε το εμπόριο. Περισσότερες εταιρείες, ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, περισσότερες περιοχές μέσα στις χώρες μας και περισσότεροι κλάδοι που θα συμμετέχουν στην διαδικασία της παγκοσμιοποίησης. Οι προκλήσεις είναι τεράστιες και ένα μεγάλο κομμάτι των λύσεων βρίσκεται μεν στις εμπορικές συμφωνίες, αλλά πολύ συχνά βρίσκεται και στην εσωτερική διάρθρωση κάθε χώρας, πώς χρηματοδοτούνται για παράδειγμα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πώς ενημερώνονται κλπ. Οι συμφωνίες ε, ελεύθερων ε, συναλλαγών ε, πολύ συχνά δεν χρησιμοποιούνται σε όλο τους το δυναμικό γιατί είτε υπάρχει άγνοια είτε δεν υπάρχουν επαρκή μέσα. Χρειάζεται λοιπόν να δουλέψουμε σε αυτό. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να συνδεθούν με τις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις έτσι ώστε να εξάγουν όχι άμεσα αλλά ενδεχομένως έμεσα. Και δεν είναι απλή διαδικασία γιατί δεν δίνονται επαρκή κίνητρα στις, μικρομεσ... στις ε, πολυεθνικές επιχειρήσεις να εντάξουν στις δραστηριότητες τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει να δημιουργηθούν δίκτυα, να την χάνουν σεβασμούς πνευματική διοκτησία, ε, να έχουν ε, κίνητρο να τη μεταφέρουν, να την παραχωρήσουν και να εντάξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις παραγωγικές αλυσίες, οι οποίες είναι πολύ περίπλοκες. Τόσο ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο. Πρέπει να προχωρήσουμε και εκεί. Όμως, αν ταυτόχρονα δεν ε, συνεργαστούμε σε ρυθμιστικό επίπεδο. Στην ε, αμοιβαία αναγνώριση των προτύπων μας δεν θα τα καταφέρουμε ούτε στο ψηφιακό εμπόριο, διότι δεν θα καταφέρουν να εξάγουν οι επιχειρήσεις. το θέμα αυτό συνδέεται και με το περιβάλλον. Όλο και περισσότερο θα υποχρονόμαστε να σεβόμαστε ε, όλο και περισσότερους κανόνες. Ε, πρέπει να βάλουμε, να χαλιναγωγήσουμε αυτό το φαινόμενο προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λοιπόν, υπάρχουν οι συμφωνίες, υπάρχουν οι εσωτερικές μεταρρυθμίσεις που να γίνουν και υπάρχει και η ευρύτερη συνεργασία ε, που ειδικά εντός της Λατινικής Αμερικής είναι σημαντικό να ενταθεί ε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υποφεληθούμε από την εμπειρία των ευρωπαϊκών χωρών. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μαρία Γκαρσία έχει το, λόγο. Thank Για το θέμα των κεφαλαίων εμπορίου και βιωσιμότητας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 Τέλεια, πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε. Και για ένα λεπτό τώρα η κυρία Έντιτα Χάρντα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Όπως είπα και στην αρχική μου παρέμβαση, ισχύει όντως ότι οι συμφωνίες αυτές είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες. Και ακριβώς επειδή ουσιαστικά είναι συμφωνίες, παγκόσμιες συμφωνίες σύνδεσης, έχουν πολλά διαφορετικά τμήματα. Εσείς συζητάτε εδώ κυρίως το εμπορικό τμήμα, το εμπορικό σκέλος. Πρέπει να σας πω όμως ότι υπάρχει και το σκέλος εκείνο, το οποίο έχει να κάνει με την πολιτική συνεργασία και το οποίο εσείς δεν συζητάτε αυτή τη στιγμή. Τα τμήματα δηλαδή εκείνα τα οποία τελούν ακόμα υπό διαπραγμάτευση, υπάρχουν τα μεικτά τμήματα εκείνα της συμφωνίας, τα οποία δεν τα έχουμε δει ακόμα. Πάντως, ε, σε κάθε μία από αυτές τις ε, τρεις συμφωνίες, ε, ένα σημαντικό τμήμα είναι τα δικαιώματα των γυναικών. Σε όλες τις συμφωνίες έχουμε και ένα εξίσου σημαντικό τμήμα μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έχουμε βέβαια και ένα κεφάλαιο που έχει να κάνει με όλα τα κοινωνικά ζητήματα τα οποία αναφέρατε και τα ζητήματα της ψηφιακής οικονομίας. Όσον αφορά τη συμφωνία με το Μερκοσούρα, δεν έχουμε νέα εντολή, διαπραγματευόμαστε ακόμα με την παλαιά εντολή. Ωστόσο, θα έλεγα ότι όλα τα τμήματα και τα δύο τμήματα είναι ιδιαίτερα καινοτόμα. Ακόμα και με την παλιά εντολή μπορούμε να συμπεριλάβουμε νέα κεφάλαια. μη φοβάστε λοιπόν ότι η τελική συμφωνία θα είναι πεπερασμένη. Θεωρώ ότι ε, μπορούμε πραγματικά να πετύχουμε πολύ περισσότερα πράγματα στο τμήμα εκείνο το οποίο δεν είναι το εμπορικό, δεν είναι το αμυγό εμπορικό. Είναι το τμήμα εκείνο στο οποίο μπορούμε να συμπεριλάβουμε, αν θέλετε, τα πιο καινοτόμα στοιχεία τη συμφωνία. Υπάρχει κεφάλαιο λοιπόν για τα δικαιώματα των γυναικών, κεφάλαιο για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και ένα κεφάλαιο που καλύπτει όλα τα ψηφιακά ζητήματα. Σα ευχαριστώ. Πρόεδρο, σα ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώθηκε κατά αυτόν τον τρόπο το πρώτο πάνελ που είχε να κάνει με τον εξυγχρονισμό των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων με τι χώρε Λατινικής Αμερικής. Ας περάσουμε τώρα στην εφαρμογή των υφιστάμενων εμπορικών συμφωνιών με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Και θα μπορούσαμε εδώ πέρα να εξετάσουμε και κάποιες πτυχές ε, του πρώτου πάνελ, στα πλαίσια της διαδικασίας εφαρμογής δηλαδή. Ο πρώτος ομιλητής είναι ο Ματίας Γιόργενσεν, προϊστάμενος του Τμήματος Λατινικής Αμερικής από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου τον καλό να πάρει το λόγο για 5 με 8 το πολύ λεπτά. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να τηρήσω το χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε στην κορασή σας. Παίρνετε πραγματικά σε μια κρίσιμη στιγμή των διμερών επενδυτικών και εμπορικών σχέσεων με τις χώρες Λατινικής Αμερικής. Ζήτημα το οποίο πραγματικά αφορά και όλο τον κόσμο όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν όλο και, περιό... όλο και περισσότερες αναδυόμενες προστατευτικές στάσεις στην περιοχή του Ατλαντικού αλλά και παγκοσμίω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα εμεί να τονίσουμε τι ισχυρέ ε, διμερεί μα σχέσει και μέσω των σημαντικών αυτών διμερών εμπορικών δεσμών να στείλουμε και ένα χειρό μήνυμα προ τα έξω προς το εμπόριο το οποίο θα πρέπει να βασίζεται σε κανόνες, προς ένα σωστό εμπορικό πλαίσιο και ένα σωστό πλαίσιο χρηστής ε, οικονομικής διακυβέρνησης. Α ασχοληθούμε τώρα λίγο περισσότερο με το συγκεκριμένο μα ζήτημα, εφαρμογή δηλαδή των συμφωνιών αυτών των εμπορικών με τι χώρε της Λατινικής Αμερικής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και το ζήτημα αυτό. Και θα πρέπει όχι απλώ να διαπραγματευόμαστε συμφωνίε, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να τι εφαρμόζουμε στη συνέχεια. Αυτό αποτελεί ουσιαστικό τμήμα λοιπόν των προτεραιοτήτων που έχουμε τη Λατινική Αμερική και δεδομένου το ότι η Λατινική Αμερική είναι η περιφέρεια εκείνη του κόσμου που έχουμε συμφωνίες μιας ευρείας γάμας ε, και παλιότερες τις οποίες όπως ακούσαμε εξυγχρονίζουμε τώρα και ελπίζω ότι βρισκόμαστε στα τελευταία στάδια της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων με όλες αυτές τις εκκρεμείς συμφωνίες. Θα ήθελα λοιπόν να πω τρία σημαντικά ζητήματα, να καλύψω τρία σημαντικά ζητήματα. Τι κάνουμε, τι θέλουμε να πετύχουμε και τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Ποια είναι τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε πετύχει. Λοιπόν, Ποια είναι η μέθοδος εργασίας. Ακολουθούμε μία εταιρική οικονομική σχέση. Προφανώς η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου εμπλέκεται άμεσα, αλλά συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη, συνεργαζόμαστε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουμε δίκτυα με επιχειρήσεις, έχουμε έναν διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και έπειτα έχουμε και εταιρικέ σχέσεις πρόσβασης στην αγορά με κράτη-μέλη και με επιχειρήσεις. Συνεργαζόμαστε μέσω των αντιπροσωπιών μας, δεν εργαζόμαστε λοιπόν σε ένα κενό. Προσπαθούμε να δείξουμε επίση και το τι κάνουμε σε εσά, υποβάλλοντάς σας εκθέσεις Ξέρετε ότι ε, στις 26 Ιουνίου θα υπάρχει και μία νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξάλληψη των εμπορικών φραγμών και θα δείτε εκεί πέρα πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε και να καταρρύψουμε τους φραγμού αυτούς και τα δύο βασικά μηνύματα εδώ πέρα είναι ότι αυξάνεται ο προστατευτισμό και ότι ε, η πρόσβαση στι αγορέ τελικά καταρρύπτει τους εμπορικούς φραγμούς. Επίσης, υπάρχει και η ε, έκθεση εφαρμογής των Συμφωνιών Ελευθεριών Συναλλαγών 2018 που θα δημοσιευθεί το Νοέμβριο. Είναι η δεύτερη φορά που υποβάλλουμε μια τέτοια έκθεση και θα καλύψουμε στην έκθεση αυτή την εφαρμογή όλων των εμπορικών συμφωνιών που έχουμε συνάψει. Τώρα, τι θέλουμε να πετύχουμε, ιδίω σε σχέση με τις χώρες Λατινικής Αμερικής. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να διασφαλίσουμε πρόσβαση στις αγορές υπηρεσιών και δημόσιων συμβάσεων και θέλουμε επίσης να εφαρμόσουμε συγκεκριμένους κανόνες για τις συμφωνίες που έχουμε με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, ιδιαίτερα ευρύες συμφωνίες. Επίσης προωθούμε τις βασικές μας αρχές στις συμφωνίες αυτές και επίσης ε, ασχολούμεθα όλους ιδιαιτέρως με το ζήτημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όλα αυτά αποτελούν επίσης και μια νέα πτυχή στον εξυγχρονισμό της συμφωνίας με το Μεξικό. Το πρώτο ζήτημα το οποίο θα ήθελα να λύσω λίγο περισσότερο, πρόσβαση στην αγορά. Προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντική πρόσβαση στην αγορά. Προφανώς αυτό ενδιαφέρει ιδιαίτερα τα κράτη-μέλη και προφανώ ενδιαφέρει επίση και του οικονομικού φορεί και τι επιχειρήσει. Ζωτικότατο λοιπόν το ζήτημα αυτό και αν δείτε τι εφαρμοστικέ εκθέσει των Συμφωνιών Ελεύθερων Συναλλαγών με την κοινότητα των Άνδεων, εκεί πραγματικά έχουμε καταφέρει να επιλύσουμε πάρα πολλά προβλήματα πρόσβαση στην αγορά, να καταρρύψουμε διάφορου εμπορικού φραγμού και εμπόδια και έχουμε καλύψει ζητήματα όπω οι ε, γεωγραφικέ ενδείξει, τα δικαιώματα διονυτική ιδιοκτησία και το σα είπα, υπάρχει και το ζήτημα των ε, αξιών, των βασικών μας αρχών. Θέλουμε βιώσιμη ανάπτυξη, κάτι το οποίο το προωθούμε πάρα πολύ. Στις συμφωνίες που έχουμε με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής και με την Κολομβία, βρισκόμαστε στη δεύτερη και τρίτη συμφωνία με τις χώρες αυτές. Είναι συμφωνίες οι οποίες εμπεριέχουν πλέον και 15 επιμέρους ε, σημεία 15 σημεία που έχουν να κάνουν με την ενίσχυση της εφαρμογής της βιώσιμης ανάπτυξης και αυτό είναι κάτι το οποίο θα παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυς με τις ε, Στι συζητήσει, μάλλον που θα έχουμε με χώρε όπω το Περού και ο Ισημερινό. Θέλουμε δηλαδή και συμφωνίε που έχουμε με τι χώρε αυτέ να προωθήσουμε τα ζητήματα αυτά, όπω η βιώσιμη ανάπτυξη. Και προωθούμε βέβαια και κάποιες βασικές μας αρχές, όπως για παράδειγμα η καταπολέμηση της διαφθοράς. Αυτό το έχουμε εντάξει, ενσωματώσει στη συμφωνία με το Μεξικό και θέλουμε να το κάνουμε και για τη Χιλή. Επίσης, ε, ε, έχουμε καινοτομήσει πάρα πολύ στις εμπορικές προτεραιότητες που έχουμε με τη Χιλή και προσπαθούμε να έχουμε καλύτερους κανόνες όσον αφορά την παγκόσμια διακυβέρνηση, να υπάρχει ε, ένα σύστημα διαιτησίας και επίλυσης διαφορών μέσω ενός επενδυτικού δικαστηρίου. Είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να περάσουμε στις περισσότερες από τις συμφωνίες αυτές. Θα μπορούσα λίγο αργότερα να μιλήσω με περισσότερες λεπτομέρειες για τις μικροσμεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα, τα αποτελέσματά μας. Σαφώς καταλήγουμε σε θετικά αποτελέσματα. Με τη Χίλη έχουμε διπλασιάσει τις εμπορικές συναλλαγές από τότε υπάρχει να ισχύει η Συμφωνία του 2002. Τριπλασιάσαμε τις συναλλαγές μας με το Μεξικό, με τις χώρες Κεντρικής Αμερικής Περού και Κολομβία. Όντω δεν έχει αυξηθεί πάρα πολύ το εμπόριο, αλλά ήδη από τι εκθέσει βλέπουμε ότι έχει διαφοροποιηθεί το εμπόριο και υπάρχουν πλέον πολύ περισσότεροι οικονομικοί φορεί που συμμετέχουν και ιδίω μικρομεσαίε επιχειρήσει από τι χώρε αυτέ. Και επί όσον αφορά τον Ισημερινό, πολύ καλό παράδειγμα αυτό το 2017 αυξήθηκε πάνω από 20% το διμερές εμπόριο. Συνοψίζοντας λοιπόν θα έλεγα το εξής. Έχουμε πολύ ισχυρέ εμπορικέ και επενδυτικέ σχέσει με την περιοχή τη Λατινική Αμερική. Παρότι ισχύει αυτό, υπάρχει ένα περιθώριο βελτίωση και ένα περιθώριο καλύτερη εφαρμογή των συμφωνιών. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η συμφωνία με το Μερκοσούρ, γιατί αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 50% του ΑΕΠ τη Λατινική Αμερική και περίπου στο 50% του δικού μα του εμπορίου. Είμαστε ιδιαίτερα φιλόδοξοι. Έχουμε ένα εκτεταμένο δίκτυο συμφωνιών, πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περιφέρεια στον κόσμο, αλλά θέλουμε ακόμα περισσότερα και θα πρέπει βέβαια να διασφαλίσουμε την ορθή εφαρμογή αυτών των συμφωνιών, γιατί μόνο αν εφαρμόζονται σωστά θα επιφέρουν ωφέλη στου πολίτε, στου καταναλωτέ και εν γέννη στο κοινό. Και αν δεν το διασφαλίσουμε αυτό, τότε πραγματικά δεν θα έχουμε την υποστήριξη, τη δημοκρατική υποστήριξη που περιμένουμε από την ευρωπαϊκή κοινωνία. Ωραία, άρα εξετάζουμε όλο και περισσότερο τη σωστή εφαρμογή των ε, συμφωνιών ε, Ελευθέρωση αλλαγών. Η κυρία Μαρία Σόρ είναι διευθύντρια στη διεύθυνση επιχειρήσεων ε, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Τιμή μου που είμαι εδώ και χαρά μου. Ονομάζομαι Μαρία Σόμπαραγκάν. Είμαι υπεύθυνη για τον ε, δραστηριότητα δανεισμού τη Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα στην Αφρική, την Καραβική και τον Ειρηνικό. Οπότε έχω και την Ασία και την, ε, ε, και την Λατινική Αμερική. Και την Καραβική, βέβαια. Είναι τράπεζε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 90% τη χρηματοδότηση μα είναι εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, το 10% εκτό. Αυτό το 10% ανέρχεται στα 8 δισεκατομμύρια, 8 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ε, ε, μοχλεύουμε επενδύσεις 25 δισεκατομμυρίων ευρώ εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε χρόνο. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ κάθε χρόνο πηγαίνει ως ε, χορηγήσεις στη Λατινική Αμερική. Ένα δισεκατομμύριο κατέτος ε, που ε, μοχλεύουν 3 με 4 δισεκατομμύρια επενδύσεων το χρόνο. Αυτό γίνεται για να ενισχύσουμε τους δεσμούς με την Λατινική Αμερική. Ε, τέσσερις είναι οι στόχοι μα που έλαβαν υπόψη, οι στόχοι, οι στόχοι του, της βιώσιμης ανάπτυξης, ένα, κλιματική δράση, δύο, ε, και ο μετριασμός και η προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές, τρίτον, οι ευρωπαϊκές προτεραιότητες και ανάλογα με την περιοχή στην οποία μιλάμε μπορεί να είναι μετανάστευση ας πούμε αυτή τη στιγμή, αλλά στην Λατινική Αμερική είναι οι δεσμοί και το να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παρούσα στη Λατινική Αμερική. Και στις επαφές μου με τους υπουργού στη Λατινική Αμερική βλέπω ότι ενδιαφέρονται πάρα πολύ για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επηρεάζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες προφανώς. Σήμερα έχουμε όπως αναφέρθηκε μεγάλη επιρροή και της Κίνας, αλλά βλέπουν ότι μοιράζονται πολλές αξίες μαζί μας και θέλουν ε, να ενισχύσουν τους δεσμούς μας. Και τέταρτος παράγοντας, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Διπλωματία. Ε, διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, αλλά και πάρα πολύ κοινέ αξίες. Δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, ε, κοινέ αρχές, κοινέ αξίες, κοινά πρότυπα τρία τα χαρακτηριστικά της ενίσχυσής μας, της βοηθειάς μας. Ε, πρώτον, αναλύουμε πολύ βαθιά τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ε, πτυχές ε, του κάθε και εδώ στις κοινωνικές πτυχές έχουμε το θέμα του φύλου. Θα, είχα, θα ήθελα να είχα χρόνο να σας πω περισσότερα, αλλά η έμφυλη διάσταση είναι πολύ σημαντική. Δεύτερον, το θέμα των προμηθειών. Εφαρμόζουμε τους ευρωπαϊκούς νόμους και κανόνες, αρχές ε, για τις κρατικές ε, προμήθειες σε κάθε ε, project που χρηματοδοτούμε, δηλαδή οι ευρωπαϊκές εταιρείες πάντοτε έχουν πρόσβαση μέσω ενός διεθνούς ανταγωνιστικού, μέσω μιας διεθνούς ανταγωνιστής δημοπράτησης διαγωνισμού. Και τρίτη, τρίτο χαρακτηριστικό ε, είναι η μόχλευση, ε, δηλαδή η κινητοποίηση και τρίτων ε, που χρηματοδοτούν επίσης τα ίδια σχέδια. Θέλουμε πάρα πολύ συγκεκριμένοι για το τι κάνουμε. Πάντα στη συμφωνία με την Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών Ευρωπαϊκής Ένωσης Λατινικής Αμερικής. με την Κολομβία και την κοινότητα των Γονάντεων. Στην Κολομβία συγκεντρώνουμε το δανεισμό μας σε δύο πράγματα. Πρώτον, η ειρνευτική διαδικασία. Η υπηρεσία εξωτερική δράση ε, μα το ζήτησε, δεδομένου ότι είμαστε Ευρωπαϊκή Τράπεζα, ακολουθούμε αυτή τη σύσταση και συνεργαζόμαστε με ένα αριθμό φόρεων στην Κολομβία για να χρηματοδοτήσουμε παραγωγικές εταιρείε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις ε, περιοχέ που είχαν πληγεί από, τον, ε, από τη από την πολεμική σύραξη. Συνολικό ποσό 400 εκατομμύρια ευρώ. Αυτές είναι οι που έχουμε αναλάβει. Επίσης, ε, μετρό της Μποκοτά, ένα από τα πιο σημαντικά ε, έργα υποδομής που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Κολομβία. Ε, ήδη εμπλέκονται ευρωπαϊκές εταιρείες και μέσω της τράπεζάς μας όλες οι εταιρείες αυτές οι ευρωπαϊκές έχουν την ίδια πρόσβαση με οποιαδήποτε άλλη. Δεν είναι ευρωπαϊκή, ε, δεν μας δίνουν κάποια προτίμηση, δεν υπάρχει κάποιο προτιμησιακό καθεστώς για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, απλά ισότιμο καθεστώς. Περού. Πέρσι δανείσαμε 150 εκατομμύρια ευρώ για ενεργειακά project ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ε, από ε, ευρωπαϊκή εταιρεία σε ό,τι αφορά την εμπειρογνωμοσύνη, την τεχνογνωσία δηλαδή ε, και τον εξοπλισμό ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που προφανώς είναι και σημαντική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί οι ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν τεχνο, ε, τεχνογνωσία που τη μοιράζονται σε όλο, με όλο τον κόσμο. Μεξικό. έχουμε μια σειρά ανοιχτών γραμμών πιστώσεως, πάντο, πιστοτικών γραμμών, πάντοτε σε σχέση με, το, με την κλιματική δράση για τη μείωση των εκπομπών πάντοτε ε, αερίων στην ατμόσφαιρα. Στηρίζουμε και εδώ ευρωπαϊκές εταιρείες, ευνελιακά project στο Μεξικό και πρόσφατα μετά την ε, Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ξεκινήσαμε μια χρηματοδότηση για την ε, διεθνοποίηση της δραστηριότητας μικρομεσαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Το συζητήσαμε και σήμερα και για ε, ευρωπαϊκές μικρομεσαίε επιχειρήσεις προφανώς που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στο Μεξικό αλλά και για μεξικανικές μικρομεσαίε επιχειρήσεις ε, που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσω χρηματοδότηση λοιπόν προωθούμε και τους στόχου των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών. Στο Μεξικό επίση συνεργαζόμαστε με τοπικέ τράπεζε για την έκδοση ομολόγων σχετικών με του στόχου ε, τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μερκοσούρ. Δεν έχω και πολύ χρόνο. κατόπιν ε, συστάσεων της Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων έχουμε ετοιμάσει ένα pipeline από project, δύο στην Αργεντινή πιο πρόσφατα, ε, ένα από αυτά ε, που αφορά την διαχείριση στερών αποβλήτων, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, με δωρεάν βοήθεια και της Ευρωπαϊκής όχι μόνο με δανεισμό. Ε, συνδυάζουμε λοιπόν διάφορες πηγές χρηματοδότησης. Στην Αργεντινή επίσης ε, συνεργαζόμαστε σε σχέδιο για το Ρίο Σαλάδο, για ένα μετρό ε, και για ηλιακά πάνελ. Βραζιλία, έχουμε χρηματοδότηση σε προγράμματα ανενώσιμων πηγών ενέργειας και πολύ πιθανώς θα χρηματοδοτήσουμε και το μετρό του Σάο Πάολο και πάλι με ε, διευκόλυνση της πρόσβασης ευρωπαϊκών εταιριών. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πάντοτε εργάζεται με βάση εντολές από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επί τη βάση αυτής της εντολής δραστηριοποιούμεθα σε αυτές τις περιοχές πάντοτε για να στηρίξουμε τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στις περιφέρειες αυτές. Ευχαριστώ. So, of... Πολύ ωραία. Αυτές είναι οι δραστηριότητες της ε, Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Επενδύσεων στη Λατινική Αμερική. Είναι η εφαρμογή λοιπόν. Και τώρα μας ενδιαφέρει η, λειτουργία των προδιαγραφών για τους εργαζομένους. Ιδιαίτερα για την Κολομβία ήταν ένα μεγάλο θέμα αυτό. Οπότε να ακούσουμε τον κύριο Ράθιο Γκίντο που είναι επικεφαλής του Τμήματος Εφαρμογής Εργασιακών Προδιαγραφών του Διεθνές Γραφείου Εργασίας. Ευχαριστώ που δώσατε τον λόγο. Ε, σας ευχαριστώ ε, που μας επιτρέπετε να σας δώσουμε την άποψη του Οργανισμού Εργασίας, του Παγκοσμίου Οργανισμού Εργασίας, του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Θα ασχοληθώ με τη Σύμβαση 169 και άλλες συμβάσεις, ιδιαίτερα για πέντε χώρες. Γιατί αυτές οι πέντε χώρες, Κολομβία, Περού, Γουατουμάλα, Σαλβαδόρ και Ονδούρας. Γιατί ο διάλογος που έχουν με τις ε, εποπτικές αρχές και τα μέτρα που έχουν ληφθεί και που θα ληφθούν ακόμη σε αυτές τις χώρες για να εφαρμοστούν οι διεθνείς εμπορικές προδιαγραφές είναι πολύ ανεπτυγμένοι. Στην ε, Κολομβία εδώ και πάνω από 20 χρόνια οι εποπτικές μας αρχές ασχολούνται με τα θέματα δημοσίων ελευθεριών, τις δολοφονίες συνδικαλιστών και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Έχουν μειωθεί όμω οι δολοφονίε αυτές τα τελευταία δέκα χρόνια. Και χαιρετίζουμε την ε, ειρηνευτική συμφωνία που υπεγράφει. Υπάρχουν κάποια νομοθετικά θέματα που πρέπει να επιληθούν. Το δικαίωμα στην απεργία και η σημασία της ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου στη χώρα για να αντιμετωπίζονται ε, διαφορές. Το έχω σημειώσει αυτό οι υποπτικές αρχές. Επίσης, ε, έχουν ληφθεί μέτρα και έχουν παρασχεθεί περισσότεροι πόροι στη, στο σώμα επιθεωρητών. Είχαμε κάνει και προτάσεις ε, πρωτότυπες για να υπάρχουν κινητά γραφεία για μακρινές περιοχές, δυσπρόσιτες. Τώρα το Περού. Υπάρχουν θέματα με το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε και τις λογικές διαπραγματεύσεις. Ορισμένες κατηγορίες ε, δεν έχουν αυτές τις δυνατότητες. Υπάρχει η τέταρτη σύμβαση εργασίας. Μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων μας είχε ζητήσει να ληφθούν μέτρα για να συμπληρώσουν την εθνική νομοθεσία για να υπάρξουν και ποινικέ κυρώσει για την καταναγκαστική εργασία. Αυτό έγινε το 2017 με μια μεταρρύθμιση του ποινικού κώδικα για να ποινικοποιηθούν ορισμένες τέτοιες εργασίες. Τώρα, Γουατεμάλα. Ότι υπήρξε μια προσφυγή κατά της χώρας αυτής για παραβίαση του δικαιώματος συνεταιρίζεστε με βάση το άρθρο 26. Είναι η πιο σημαντική δυνατότητα που έχει ο οργανισμός μας για παραβιάσεις των συμβάσεων του ILO. Και με βάση τη διαδικασία μπορεί να δημιουργηθεί και μια επιτροπή έρευνας όμως ε, έχουν ληφθεί διάφορα μέτρα και υπεγράφει μια τριμερή συμφωνία τον περασμένο Νοέμβριο για να εφαρμοστεί ένα οδικό χάρτη που υπεγράφει το 2015 με συγκεκριμένα μέτρα που προέβλεψε η κυβέρνηση για να γίνεται πλήρω σεβαστή το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε. Και υπάρχει και μία επιτροπή για την επίλυση συγκρούσεων Βέβαια στην Γουατεμάλα δεν λειτουργεί τόσο καλά όσο στην Κολομβία. Και τώρα αποφασίστηκε να υπάρξει μια νέα τριμερής επιτροπή για τις εργασιακές σχέσεις και το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε που ε, θα ασχοληθεί με όλα τα θέματα που έχουν φυγεί. Όμως οι προδιαγραφές μας έχουν ληφθεί υπόψη για να γίνονται περισσότερες επιθεωρήσεις εργασίας και ενεκρίθη ένας νέος νόμος που επιτρέπουν στους επιθεωρητές να επιβάλλουν πρόστιμα. Παλιά δεν γινόταν αυτό. Κάποιο άλλο σώμα με το οποίο ασχολούμεθα τακτικά είναι το Ελσαλβαδόρ. Δεν υπάρχει αποτελεσματικός κοινωνικός διάλογος σε αυτή τη χώρα και το έχουμε τονίσει επανειλημμένα. Πρέπει να ε, επανενεργοποιηθεί μια επιτροπή διαλόγου για εργατικά θέματα, γιατί υπάρχουν θέματα παιδικής εργασίας, καταναγκαστικής εργασίας και του δικαιώματος ε, δημιουργίας ε, εργατικών ενώσεων. Και με τις ε, Ονδούρες έχουμε ασχοληθεί επανειλημμένα. για την εφαρμογή συγκεκριμένα τη σύμβαση 87 που αφορά σοβαρές παραβιάσει συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Έχουν γίνει εγκλήματα κατά συνδικαλιστών, αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι ότι το 2016 επίσης ζήτησαμε την εφαρμογή της Σύμβασης 169 για τους γηγενεί πληθυσμούς. Η κυβέρνηση έλαβε ταχύτατα μέτρα, ενεκρίθηκε ένα νόμο για τη διαδικασία διαβούλευση με του γηγενεί και για την επιθεώρηση εργασίας θα προωθήσουν ένα νέο νόμο μετά την συζήτηση που έγινε σε μια συνδιάσκεψή μας. Παρόμοια προβλήματα υπάρχουν και σε άλλες χώρες της περιοχής. Την Κεντρική Αμερική, την Κολομβία και το Περού. Υπάρχουν επίπεδα βίας που ποικίλουν, αλλά η Γουατεμάλα, η Ονδούρας και η Σαλβαδόρα παρατηρούμε προβλήματα βίας κατά συνδικαλιστών. Χρειάζονται και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις για να υπάρχει πλήρης δυνατότητα λειτουργίας εργατικών ενώσεων και συλλογικών διαπραγματεύσεων. Πρέπει να καταπολεμηθεί η παιδική και εργασία στις χώρες αυτές. Όλες πρέπει να ενισχύσουν τις επιθεωρήσεις εργασίας και να ενισχύσουν τον κοινωνικό διάλογο. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή μια ενοποιημένη αντίληψη για την εφαρμογή των διεθνών προδιαγραφών εργασίας. Τώρα, τι δράσεις έχουν αναλυφθεί από την υπηρεσία, το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Χάρη και στη βοήθεια που μας δίνει η Γενική Διεύθυνση Trade και Αντεύκο. Μας επιτρέπουν να εργαστούμε με φορείς των χωρών αυτών, ιδιαίτερα για τον κοινωνικό διάλογο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κάποια βελτίωση, αλλά πολλά ακόμη έχουμε να κάνουμε. Και βεβαίως και η κοινωνία των πολιτών πρέπει να εμπλέκεται περισσότερο στις εμπορικές μας συμφωνίες έχουμε το λεγόμενο DAC τα, τα λεγόμενα εθνικά συμβουλευτικά συμβούλια οι ομάδες που είναι αρμόδια συγκεκριμένα για την εφαρμογή των κεφαλαίων για το εμπόριο και τη βιωσιμότητα. Υπάρχουν αυτά τα περίφημα 15 σημεία από την Επιτροπή που θα έπρεπε να είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή. Και ο πρόεδρος ε, της EU-DAC για την Κολομβία, το Περί, το Εκουαδόρ είναι ο Τζουζέπε Τζουλιάνο. Και εδώ στο λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Νομίζω ότι μπορώ να μιλήσω την όμορφη μητρική μου γλώσσα, τεταλικά. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί έτσι μου δίνεται και ευκαιρία να σας εξηγήσω λίγο μέσω της παρέμβασής μου αυτής πώς συμμετέχει όντως η κοινωνία των πολιτών σε αυτές τις συμφωνίες. Μιλάμε λοιπόν για εγχώριες συμβουλευτικές ομάδες οι οποίες ασχολούνται με την παρακολούθηση της εφαρμογής των συμφωνιών αυτών. Και εδώ πέρα αναφερόμαστε κυρίω στη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με την Κολομβία, το Περού και τον Ισημερινό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώ τελικά η κοινωνία των πολιτών, για παράδειγμα οι οργανώσει επιχειρηματιών, οι οργανώσει των εργαζομένων, η ενός των καταναλωτών, για παράδειγμα, οι περασπιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή οι ε, του περιβάλλοντο, πώς εμπλέκονται σε αυτές τις συμφωνίες. Πάρα πολλές φορές στο παρελθόν είχαν αντιδράσει έντονα λέγοντας ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλες οι ήταν ασυμμετρική μάλλον η στάση συμφωνίες αυτές ανάμεσα στις οικονομικές προτεραιότητες και τις υπόλοιπες προτεραιότητες. Και ξέρετε ότι υπήρχε, κύριε Πρόεδρε, και ένα οδικό χάρτη, στον οποίο είχα συμμετάσχει και εγώ πάρα πολύ, προκειμένου να καταφέρουμε μέσω των συμφωνιών αυτών να ξεπεράσουμε κάποια προβλήματα που υπήρχαν. Μία εφαρμογή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φαινόμενα τιμωρησία, καταπάτηση των δικαιωμάτων των συνδικαλιστών και το καθεξής. Τα τελευταία λοιπόν 34 χρόνια οι ίδιες οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που είχαν εκφράσει τέτοια αντίδραση στο παρελθόν συνειδητοποίησαν ότι όντως θα μπορούσαν μέσω των επιτροπών αυτών παρακολούθησης να έχουν και αυτές ένα λόγο. Κάποια προβλήματα τα αντιμετωπίζουμε ακόμα στο Περού, στη Κολομβία, ακόμα και στον Ισημερινό, γιατί βλέπουμε ότι εκεί πέρα ότι υπάρχουν ακόμα κυβερνήσεις οι οποίες θεωρούν ότι ε, οι επιτροπές αυτές βασικά θα πρέπει να δημιουργούνται με συμμετέχοντες από την ίδια την κυβέρνησή τους. Σε κάποιες χώρες θέλουν να βάλουν και τον ίδιο τον Υπουργό τους να συμμετέχει σε αυτές τις ε, ομάδες παρακολούθησης. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε βέβαια είναι να έχουμε απόλυτη αυτονομία και ανεξαρτησία και να μπορούμε πραγματικά να επεμβαίνουμε συμβουλεύοντας αυτές τις κυβερνήσεις. Καταφέραμε πάντως ε, να πετύχουμε αρκετέ βελτιώσει. Αυτή τη στιγμή στην Κολομβία, για παράδειγμα, έχουμε ένα DAG, μια τέτοια εγχώρια συμβουλευτική ομάδα, την οποία την έχουμε συστήσει με τη σύμφωνη γνώμη τη κυβέρνηση και όντω λειτουργεί αποτελεσματικά. Η συμφωνία με την Κολομβία, το Περού και την Ισημερινό, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώ και τι τρει αυτέ χώρε, είναι πάρα πολύ σημαντική για τη συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών. Στη συμφωνία λέγεται ότι η διαβούλευση θα γίνεται μέσω διαβούλευση εν γέννη του κοινού. Κάτι τέτοιο να φέρετε συμφωνία. Εμεί το τονίσαμε αυτό και είπαμε ότι δεν μπορούσαμε να το δεχθούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Μέσω του διαλόγου επίση που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Επιτροπή. Και καταφέραμε τελικά σιγά σιγά ερχόμενα σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία τρία χρόνια να πετύχουμε θετικά αποτελέσματα. Γιατί καταφέραμε να πετύχουμε τελικά κοινέ επιτροπέ. Δηλαδή Κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργήσαμε αυτέ τι όντω εγχώριε εσωτερικέ συμβουλευτικέ ομάδε. Δεν έχει κανένα νόημα να ακούμε την κοινωνία των πολιτών ξεχωριστά μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο στην Κολομβία, μόνο στο Περού ή μόνο στον Σημερινό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δημιουργούμε μεικτέ, κοινέ τέτοιε εγχώριε συμβουλευτικέ ομάδε. Για παράδειγμα, να έχουμε ομάδε όπου θα έχουμε συνδικαλιστέ από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνδικαλιστέ από την Κολομβία. Το ίδιο για το Περού, το ίδιο για την, τον Ισημερινό. Κατά αυτόν τον τρόπο, μέσω τη κοινή αυτή συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων μπορούμε να γνωρίζουμε ποιε είναι οι επιπτώσει τη συμφωνία, για παράδειγμα στι εισαγωγέ ή εξαγωγέ, αν υπάρχουν θετικέ ε, ή αρνητικέ επιπτώσει, ποιο είναι ο αντίκτυπο τελικά τη συμφωνία που εφαρμόζεται. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο το οποίο θέλω να τονίσω. Δεν έχουμε ακόμα μηχανισμούς επιβολής κυρώσεων. Δεν έχουμε διορθωτικούς μηχανισμούς πραγματικούς. Και παρόλα αυτά, εμείς παρουσιάσαμε τα προβληματικά αυτά σημεία στην κυβέρνηση του Περού και καταφέραμε τελικά ερχόμενοι σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές της κυβέρνησης μέσω των μεικτών αυτών συμβουλευτικών ομάδων να τονίσουμε ότι όντως υπήρχαν σημαντικές αντιφάσεις στη συμφωνία αυτή και το ότι η εφαρμογή τελικά της συμφωνίας γινόταν με τέτοιο τρόπο που τελικά δεν τηρούνταν τα δικαιώματα όλων αυτών που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να συμμετέχουν σε αυτές τις συμφωνίες. Και μάλιστα η ίδια η Επίτροπος Μάλστρομ ζήτησε από τις αρχές του Περού να ανταποκριθεί στα αιτήματα τα οποία εμείς υποβάλαμε. Είδαμε λοιπόν ότι υπήρχαν σημαντικά κενά, σημαντικές αδυναμίες στη συμφωνία με το Περού και περιμένουμε ακόμα την απάντηση της περουβιανής κυβέρνησης. Ακόμα και το Κοινοβούλιο της Καταλωνίας περιμένει ακόμα την απάντηση από την κυβέρνηση του Περού. Και το πετύχαμε αυτό ακριβώς επειδή συμμετέχει έντονα η κοινωνία των πολιτών τονίζουμε τα κακό κείμενα και θεωρούμε ότι θα καταφέρουμε να έχουμε από τις αρμόδιες αρχές του Περού μια διόρθωση των πτυχών εκείνων της συμφωνίας που είναι προβληματικές. Για τον Ισημερινό τώρα θα έχουμε μια συνεδρίαση κοινή της κοινωνίας των πολιτών, δηλαδή από την Κολομβία, το Περού και τον Ισημερινό και από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουμε συμμετοχή σε μια μεικτή χώρια συμβουλευτική ομάδα. Να κάνω επίσης μια γενική παρατήρηση που είναι κάτι το οποίο με έχει απασχολήσει στα πλαίσια της σημερινής συζήτησης. Το γενικό αυτό πλαίσιο που έχουμε, προστατευτισμός, λαϊκισμός, οι αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης και το καθεξής. Η Λατινική Αμερική είναι πραγματικά η ήπειρος με την οποία μπορεί να συνεργαστεί να συνασπιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και να δημιουργήσει ένα τέτοιο εμπορικό σύστημα. Γιατί στη Λατινική Αμερική οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έχουν ήδη έναν εργατικό κώδικα ο οποίος είναι πάρα πολύ παλιός, ήδη από την δεκαετία του 80 και του 90 είχαν καταφέρει να προχωρήσουν σε απαραίτητες εργατικές μεταρρυθμίσεις, ακολουθώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν οργανώσει την κοινωνία των πολιτών τους πάνω στο ευρωπαϊκό μοντέλο. Το Μερκοσούρα αυτή τη στιγμή αποτελεί ένα φόρουμ στο οποίο συμμετέχουν πέρα από τους οικονομικούς φορείς και πάρα πολλοί εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Και ακριβώς επειδή ε, τα ισπανικά και τα πορτογαλικά είναι επίσημες ε, γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προφανώς είναι γλώσσες που μιλούνται πάρα πολύ στην Εθνική Αμερική, είχαν τη δυνατότητα όλοι οι συμμετέχοντες στα φόρουμ αυτά από την πλευρά της Λατινικής Αμερικής να μελετήσουν τα κείμενα τα οποία ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει μια έντονη προστιθέμενη αξία σε αυτές ε, τις συμφωνίες. Και αυτό ισχύει και για τη Συμφωνία της Χιλής. Ας μην ξεχνάμε ότι Ξεκινήσαμε καταρχάς με συμφωνίες σύνδεσης με τις χώρες αυτές, όπου πέρα από τις εμπορικές σχέσεις προβλέπεται και η πρόθεση κάποιων βασικών αξιών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συνδιαλέγεται περισσότερο με την Εθνική Αμερική στα πλαίσια της νέας αυτής οικονομίας που αναδύεται. Παρακαλώ τώρα ερωτήσεις. Ο κύριος Φίσας, εισηγητής μας για την Κολομβία και το Περού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγχαρητήρια στους εισηγητές για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις τους. Χτες ε, έλαβε χώρα μια συνάντηση παρακολούθηση της συμφωνίας με τις χώρες των Άνδεων. Συμμετείχαν και συνδικαλιστές από τον κλάδο της ε, μπανάνας ανησύχησα πολύ διότι μου είπαν πως οι εργαζόμενοι στον κλάδο βρίσκονται σε μια κατάσταση δουλεία σχεδόν, έτσι μας το είπαν. Ε, με πολύ χαμηλούς μισθούς και με δικαιώματα ε, πολύ περιορισμένα. Έτσι μας το είπαν. Αυτό μου δημιουργεί σημαντικές ανησυχίες ε, πρώτον σε ό,τι αφορά τα ε, εργατικά τους δικαιώματα και δεύτερον διότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα κοινωνικό dumping σε σχέση με του εργαζόμενου των ευρωπαϊκών ε, επιχειρήσεων. Δηλαδή, αν οι εργαζόμενοι του σημερινού, συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και άλλων χωρών των Άντεων εργάζονται σε τέτοιου είδου συνθήκες, αυτό μπορεί να μολύνει μέσω κοινωνικού dumping ε, και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά τις εργασιακές συνθήκες που ε, παραχωρούν στους δικούς τους εργαζόμενους. Ε, θα ήθελα να ακούσω την άποψη του κυρίου Γιόργενσεν που ήταν παρόν, τι σκοπεύει να κάνει η Κομισιόν γι' αυτό και επίσης του κυρίου ε, Γκουίντο, Γκίντο, που μας μίλησε για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Τώρα μια ερώτηση στην κυρία Σο Μπαραγκάν είναι προφανώ σημαντικότατη η στήριξη που μπορεί να δοθεί ε, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, ξέρουμε ότι ε, οι μεγάλες επιχειρήσεις όπως αυτές που κατασκευάζουν το μετρό και άλλες ξέρουν που θα βρουν χρηματοδότηση. Τι γίνεται με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κυρίως με, τις, με την πληροφόρηση που πρέπει να τους δίνεται σε ό,τι αφορά τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που έχουν στη διάθεσή τους. Με την κυρία Ροδρίγε Πινιέρο το είπαμε και όταν συζητούσαμε το Μεξικό. Πολύ συχνά οι μικρομεσαίε επιχειρήσει δεν γνωρίζουν τι δυνατότητε που του δίνουν συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών. Ευχαριστώ πολύ. ΙΜΑ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγχαρητήρια και από μένα στους ομιλητές σαφέστατες και πολύ συγκεκριμένες οι παρεμβάσεις τους. Έχω τον εξή προβληματισμό να εκφράσω και μια ερώτηση. Προ τον κύριο Ματία Γιώργενσεν, θέλω να πω το εξή. Ε, νομίζω ότι είπατε πω τον Νοέμβριο ξεκίνησε μια έκθεση ε, εφαρμογή σε ό,τι αφορά τι εμπορικέ ε, συμφωνίες του 18. Ε, πού βρίσκονται, τι φιλοδοξίες έχουμε για αυτές τις μελέτες εκθέσεις. Εμείς ε, έχουμε ζητήσει διάφορα ε, πράγματα σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση. Για παράδειγμα, ε, να μπούμε σε στοιχεία τα οποία έχουν σχέση με, την εμπορική, με τις εμπορικές σχέσεις, αλλά όχι μόνο αριθμητικά. Να δούμε και ποιοτικά την εφαρμογή. Για προς την κυρία Σόμπαραγκάν θα ήθελα να πω το εξής. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση και εγώ προασπίζομαι την πολιτική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που πρέπει να βοηθάει ε, τη χρηματοδότηση προγραμμάτων. Στην Κολομβία όμως μας είπαν ότι η ε, ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν έχει δημιουργήσει ένα γραφείο επιτόπου ε, για να στηρίξει την ειρηνευτική διαδικασία. Ε, έχει ανοίξει από τότε αυτό το γραφείο ακόμα έχετε δυσκολίες. Κύριε Κίντο, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των συμβάσεων του ε, Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, Οργάνωσης Εργασίας. Εγώ στις χώρες της Λατινικής Αμερικής που επισκέφθηκα είδα ότι ορισμένες χώρες που έχουν υπογράψει την σύμβαση του 98 αλλά δεν την εφαρμόζουν, ε, δεν έχουν συλλογικές ε, συμβάσεις, ε, δεν προβλέπουν αυτό το θεσμό. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε τι μπορεί να γίνει έτσι ώστε να τις εφαρμόσουν αυτές οι συμφωνίες που έχουν υπογράψει, όπως το 98. Ο κύριος, για τον κύριο Τζουζέπη Ιουλιάνο. Στην επίσκεψή μας στο Περού και την Κολομβία, είδαμε διαφορές ανάμεσα σε αυτές τις δύο χώρες ό,τι αφορά την εφαρμογή των συμφωνιών. Επίσης διαπιστώσαμε ότι το επίπεδο ανάπτυξης της Κοινωνία των πολιτών, οριμότητα των οργανώσεων, στήριξης τη κυβέρνηση στις οργανώσεις τη Κοινωνία των πολιτών είναι διαφορετικό από τη μία χώρα στην άλλη. Είπατε κάτι με το οποίο συμφωνώ πλήρως. Η κυβέρνηση προτιμάει να χρησιμοποιεί τους κλαδικού μηχανισμούς παρακολούθηση που υπάρχουν στο ε, Υπουργείο, όμως αυτό δεν είναι αρκετό ούτε αποτελεσματικό κατά την άποψή μας. Ε, στην περίπτωση του Περού που είναι πιο άσχημη κατάσταση, κάποτε κατάλαβα στείλατε μία επιστολή, δεν ξέρω τι θα κάνετε για την Κολομβία, γιατί είναι αλήθεια πως και στις δύο περιπτώσεις δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή το εργαλείο το οποίο συμφωνήσαμε για την συμμετοχή στο διάλογο της κοινωνίας των πολιτών ανεξάρτητα αν, από το αν η πρόοδος έχει γίνει σε διαφορετικούς βαθμούς σε δύο χώρες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να αναφερθώ και πάλι στις Κυρος, στη Γουατεμάλα. Επανειλημμένα αναφέρθηκε, το είπε και η κυρία Γκαρσία. υπόθηκε ότι μια φορά μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Γουατεμάλας ε, επιχειρήθησαν κυρώσεις και δεν λειτουργήσαν. Αλλά δεν είναι αυτό απόδειξο, δεν πρέπει ποτέ να ε, επιχειρήσουμε να τις επιβάλλουμε. Πώς πρέπει να τις επιβάλλουμε, αυτό είναι το ερώτημα. Δεν πρέπει να τα παρατήσουμε τόσο γρήγορα. Δεν πρέπει απλώ να λέμε μόνο μέσω διαλόγου θα τα λύσουμε. Ξέρουμε από άλλα παραδείγματα ότι δεν αρκεί πάντα ο διάλογος. Για τις προδιαγραφές του ILO ο κύριος ε, Γουίντο μας εξήγησε πόσο δύσκολη είναι η εφαρμογή και πόσο μακροχρόνιες και χρονοβόρες οι διαδικασίες. Νομίζω ότι θα πρέπει να θέτουμε ως προϋποθέσεις τις οκτώ βασικές ε, προδιαγραφές του ILO. Αυτό θα πρέπει να είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Αυτό θα πιέσει τους εταίρους μας να τις εφαρμόσουν, να τις επικυρώσουν τάχιστα. Γιατί είναι ελάχιστες προδιαγραφές αυτές. Και αν δεν το καταφέρουμε αυτό πριν ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση, μετά είναι πολύ δύσκολο να τις επιβάλλουμε. Έχουμε και παραδείγματα. Πολλοί εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών μου είπαν ότι δεν υπάρχει διαφάνεια, δεν ενημερώνονται για το τι γίνεται, για τις προθέσεις ε, και τα εγχειρήματα της κυβέρνησης. Και αυτό δεν βοηθάει την συνεργασία φυσικά. Θα πρέπει να βρούμε τρόπο να ενισχυθεί αυτή η συνεργασία. Δεν ξέρω μήπως ορισμένοι δεν τη θέλουν ή δεν είναι συνηθισμένο στην Λατινική Αμερική να λαμβάνεται σοβαρά η κοινωνία των πολιτών. Πρέπει να τους ε, καταδείξουμε πόσο σημαντική και πόσο θα τους βοηθήσει αυτή η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Πρέπει να τους στηρίξουμε λοιπόν. Να στηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών και να δούμε και τι μέσα θα ήταν αναγκαίο τόσο ώστε να συμμετέχει και να λαμβάνεται πιο σοβαρά υπόψη η κοινωνία των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Τέσσερις ερωτήσεις από πλευρά μου. Τζουζέπε, ποια είναι η εντύπωσή σου. Πώς λειτουργούν οι οργανισμοί DAX στις ε, χώρες αυτές. Έχουν πόρους για να λειτουργήσουν. Ποια είναι η οικονομική τους κατάσταση. Μπορούν να παίξουν το ρόλο τους. Και να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ευθύνες τους. Κύριε Γκίντο, Έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των εξαγωγικών εταιριών και των υπολείπων. Οι εξαγωγικές εταιρείες αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές και να δέχονται υποχρεώσεις, ε, επιθεωρήσεις, αλλά με τις υπόλοιπες έχουμε πρόβλημα. Ισχύει αυτή η εντύπωσή μου. Κυρία Σόμπαραγκαν, βεβαίως ε, η Κίνα είναι ανταγωνιστής μας. Αλλά η Κίνα δεν έχει τόσες συμφωνίες ε, όσες εμείς. Είναι όμως μήπως πλεονέκτημα αυτό. Για την Κίνα. Γιατί η Κίνα έχει εντελώ διαφορετικέ διαδικασίε και εντελώ διαφορετικό στρατηγικό προσανατολισμό και επενδυτικό προσανατολισμό. Τι μπορούμε να κάνουμε εμεί για να αντεπεξέλθουμε σε αυτόν τον ανταγωνισμό. Και κύριε Γιώργενσεν, τι ρόλο παίζει για την εφαρμογή οι αντιπροσωπεία τη Ένωση τόπου. Γιατί είναι σημαντικό ο ρόλο του, αναμφίβολα. Υπάρχουν κάποιε κατευθύνε γραμμέ που δίδονται προ τι αντιπροσωπείε για να ξέρουν τι να κάνουν για να βοηθήσουν την εφαρμογή. Και πώς θεωρείτε ότι συνεργάζεται η Γενική Διεύθυνση Trade με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Είναι καλή συνεργασία. Είναι υποτονική. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Λοιπόν, με την αντίστροφη σειρά τώρα. Τζουζέπε, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λοιπόν, να απαντήσω στην ερώτηση που έκανε η Μακουλάδα. Ουσιαστικά είναι η ερώτηση που θέσετε και εσείς κύριε Πρόεδρε για τον πιθανό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και η διαφορά που υπάρχει από τη μία χώρα στην άλλη όσον αφορά την κοινωνία των πολιτών. Αναφερόμαστε εδώ πέρα σε ανθρώπους οι οποίοι όπως και εγώ ενδιαφέρονται πάρα πολύ για την ε, Λατινική Αμερική. Ο Χατ Πέρινγκτον και ένας ε, πολύ σημαντικός ιστορικός ε, έλεγε ότι δεν θα πρέπει να μιλάμε για μία Λατινική Αμερική, αλλά για πολλές Λατινικές Αμερικές. Αυτό ισχύει σίγουρα. Δεν μπορούμε μονομερός να βλέπουμε όλες αυτές τις χώρες. Η σχέση που έχουμε με την Κολομβία, το Περού, τον Ισημερινό, Μολονότι οι σχέσεις είναι διμερείς, ανάμεσα στις χώρες αυτές υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές. Ξέρετε ότι βιώσαμε την όλη ειρηνευτική διαδικασία του Πρόεδρου Σάντο στην Κολομβία. Ξέρετε ότι χθε έχουμε τον νέο Πρόεδρο της Κολομβίας που πρέπει και αυτός πάλι να δούμε πώς θα επηρεάσει τις ε, συμφωνίες αυτές, ε, τις ειρηνευτικές συμφωνίες, γιατί αυτό με τη σειρά του θα πειράσει και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η κυβέρνηση του Περού δεν αντέδρασε με τον ίδιο τρόπο σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε ως κοινωνία των πολιτών. Τονίζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα, ότι υπάρχουν αντιφάσεις. Δεν είναι ποτέ δυνατό να χρησιμοποιούν εγχώριες επιτροπές ε, αυτές οι χώρες. Η Κολομβία αντέδρασε σωστά, θεωρώ διασφαλίζει πλέον την αυτονομία της Εθνικής Συμβουλευτικής Ομάδας, αλλά στο Περού δυστυχώς δεν έχει γίνει ακόμα κάτι τέτοιο. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πρέπει να θίξουμε το πρόβλημα αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιληφθεί ερχόμενη σε επαφή με τους εταίρους, με τις αρμόδιες αρχές δηλαδή του Περού εν προκειμένου. Η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όντως κινητοποίησε πάρα πολλούς πόρους, 3 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να συμμετάσχει περισσότερο η κοινωνία των πολιτών, να κινητοποιηθεί η κοινωνία των πολιτών και να υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα από τη μία χώρα στην άλλη, εκεί που υπάρχουν δηλαδή πολυμερείς συμφωνίες. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να επιθυμίσω στους φίλους ευρωβουλευτές ότι εδώ η αρχή ουσιαστικά είναι κάπω λανθασμένη. Εμεί θα πρέπει να ζητούμε από τις κυβερνήσεις εταίρους Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτοί, αυτοί να εγγυηθούν και να διασφαλίσουν τα μέσα συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών σε αυτές τις επιτροπές παρακολούθησης. Όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση να το κάνει αυτό με τα δικά της τα μέσα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική αρχή. Και όντω βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει το κόστο αυτό μέχρι σήμερα. Αλλά πρέπει εμεί να επιμείνουμε προκειμένου οι κυβερνήσει των χωρών εταίρων να αναλάβουν αυτές το ρόλο αυτό, αυτές να διασφαλίσουν τη συμμετοχή της κοινωνία των πολιτών του, στις επιτροπέ παρακολούθηση. Επ' αυτού, όπως το είπα, το μόνο μπορούμε να κάνουμε εμεί είναι να τονίζουμε κάθε φορά τι αντιφάσει που υπάρχουν και τα προβλήματα που υπάρχουν και να κάνουμε ουσιαστικά καταγγελίες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά εσείς ως ευρωβουλευτές πρέπει να θέσετε την πολιτική διάσταση του προβλήματος. Εσείς ουσιαστικά μπορείτε να συμβάλλετε πιο αποτελεσματικά. Ο Ράτσιο Γκουίντο το είπε πάρα πολύ καλά αναφερόμενο στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Εσείς πραγματικά είστε αυτοί οι οποίοι προωθείτε τις αρχές τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς βασιζόμαστε πάρα πολύ στην εργασία που μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Περιμένουμε τη δική σας συμβολή. Ο κύριος Γκίντο. Ευχαριστώ πολύ. Για τις δύο πρώτες ερωτήσεις. Αυτό που έχει να κάνει με τις, ε, τις δυσχέρειες που έχουν εργαζόμενοι στο χώρο των άνδεων ε, ε, που ασχολούνται με την καλλιέργεια της μπανάνας και για την επικύρωση συμφωνιών και συμφώνων που κατόπιν δεν εφαρμόζονται. Η συνηθισμένη απάντηση. Οι εργαζόμενοι σε ορισμένου ε, κλάδους, όπως συγκεκριμένα στην καλλιέργεια της Μπανάνα, που δεν τηρούνται οι συμφωνίε στην περίπτωσή του, έχουν πρόσβαση στου μηχανισμού ελέγχου, του δικού μα, Μπορούν να υποβάλουν προσφυγέ στην Επιτροπή για τι Συνδικαλιστικέ ελευθερίε με βάση το άρθρο 24 του καταστατικού μας μπορούν να ζητήσουν να σταλούν παρατηρητές συγγνώμη όχι καλύτερα να στείλουν ε, τις διαμαρτυρίες τους ε, στα κείμεν, στις επιτροπές μας τις γνωρίζουν τις διαδικασίες αυτές στην περίπτωση της Κολομβίας χρησιμοποιούν πολύ αλλά και σε άλλες περιπτώσεις από την Κεντρική Αμερική και την ε, Βόρεια και την Νότια αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα ε, λαμβάνουμε πολλές προσφυγές από την Λατινική Αμερική είναι ο πρώτος μας πελάτης ε, η περιοχή αυτή. Αλλά οι εργαζόμενοι ζητούν συγκεκριμένες λύσεις στα προβλήματά τους. Και πολλές φορές η εξέταση ε, μιας προσφυγής μπορεί να πάρει ένα-ενάμιση χρόνο. Ενώ οι εργαζόμενοι ζητάνε να τους πληρώσουν για την εργασία τους. Εμείς βοηθήσαμε όμως, συγκεκριμένα στην Κολομβία για να υπάρχουν μηχανισμοί επίλυσης ε, εργατικών, εργασιακών διαφορών. Η Κολομβία έχει μια τέτοια επιτροπή για να αντιμετωπιστούν ε, οι προσφυγές που υποβάλλονται στον ILO. Ε, Επιλύσαμε πολλές σημαντικές πολλές προσφυγές αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς και λύσαμε πολλές εκατοντάδες Το θέμα λοιπόν είναι ανακλάδο. Πρέπει να δούμε που υπάρχουν προβλήματα. Στην περιοχή των Άνδεων έχουμε το πρόβλημα με την μπανάνα, με τα λουλούδια, με τα ορυχεία. Εκεί έχουμε τα προβλήματα. Παιδική εργασία, έλλειψη συγκαλιστική ελευθερία, χαμηλή μισθή. Και το... Ε, βέβαια, βέβαια μειώνεται η βία στην Κολομβία. Να ενισχύσουμε τι οργανώσει των εργαζομένων επιτόπου. Αυτό είναι το θέμα. Αν δεν υπάρχουν ισχυρέ και πραγματικά ανεξάρτητες τέτοιε εργατικέ ενώσει μπορούμε να επικυρώσουμε ό,τι θέλουμε. Μετά δεν θα εφαρμοστούν ούτε σε εθνικό επίπεδο, ούτε σε διεθνές. Τώρα για το Μερκοσούρ, κάτι που αξίζει τον κόπο. Οι διαφορές εργασιακέ εργασιακές σχέσεις, όπως είπε και ο συναδελφός μου εδώ, οι διαφορές είναι τεράστιες. Σε ορισμένες χώρες είναι πολύ ισχυρές και σε άλλες πολύ αδύναμες. Ενώ γίνονται εργασιακές μεταρρυθμίσεις που σε ορισμένες χώρες προχωράνε και σε άλλες όχι γιατί υπάρχουν αντιστάσεις. Με ρωτήσατε. Να επιχειρήσουμε πριν υπογραφεί μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών να επιβάλλουμε κάποιες προδιαγραφές. Εμείς δεν έχουμε να σας κάνουμε συστάσεις. πριν ή μετά λοιπόν να επιχειρήσουμε να επιβληθούν αυτές οι προδιαγραφές. Εμείς από τις υποπτικές αρχές διαπιστώνουμε ότι οι απευθυνόμενοι στον αελο αυτό που θέλουν είναι να υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση από τις κυβερνήσεις. Στο Κατάρ, τον στην Κολομβία, στη Γουατεμάλα διαπιστώθηκε αυτή η βούληση να δεσμευτούν για συγκεκριμένες δράσεις. και να εφαρμοστούν οι διεθνείς εργασιακές προδιαγραφές. Αυτό φάνηκε μέσω της εκπόνησης οδικών χαρτών με συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να ληφθούν. Και τελευταία ερώτηση, εξαγωγικές εταιρείες και μη, σε σχέση με το σεβασμό των προδιαγραφών. Αυτό που διαπιστώνουμε εμείς είναι ότι καμία επιχείρηση, είτε μικρή είτε μεγάλη, εξαγωγική ή όχι, καμία δεν θέλει να αναφέρεται στις εκθέσεις μας και στις ε, ακροάσεις μας. Όταν ε, μια χώρα είναι αντικείμενο εξέτασης από τον οργανισμό μας, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει βούληση να συμμορφωθούν με τις ε, συμβάσεις. Ανεξάρτητα από το μέγεθος και το χαρακτήρα της επιχείρησης. Ίσως είναι πολύ πιο εύκολο για κάποιες μεγάλες εταιρείες. Έχουν τους πόρους και τα τμήματα. Αλλά καμία δεν θέλει να καταγγελθεί ως επιχείρηση που δεν σέβεται τις διεθνείς εργασιακές προδιαγραφές. Αυτό διαπιστώνουμε εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Σο Μπαραγάν. Να απαντήσω στις δύο πρώτες ερωτήσεις στα ισπανικά. Σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Προφανώς η στήριξή τους είναι απαραίτητη. Είναι αυτές που δημιουργούν θέσεις εργασία. Είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στη Λατινική Αμερική και όταν συνομιλούν μαζί του ή μέσω των επιμελητή, των εμπορικών επιμελητήων, μα λένε ότι η πρόσβασή του στη χρηματοδότηση είναι το μεγαλύτερο εμπόδιό τους, το μεγαλύτερο εμπόδιο στην ανάπτυξή τους, στη μεγέθυνσή τους. Οπότε πρέπει να διευκολύνουμε τη χρηματοδότησή τους με μεγαλύτερη πρόσβαση, πιο εύκολη πρόσβαση και πιο μακροχρόνια δάνεια. Τώρα, σε σχέση με τη διεθνοποίησή τους, ε, ε, υπάρχει κι άλλος ένας παράγοντος που τις επηρεάζει που είναι η ψηφιακή μετάβαση. Το ίντερνετ των πραγμάτων, το ηλεκτρονικό εμπόριο, όλα αυτά αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν αποτελεσματικά να χρησιμοποιήσουν ή όχι τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Ένα άλλο ζήτημα ε, πράγματι, πολύ συχνά χρηματοδοτούμε μεγάλα σχέδια, αλλά πολλές φορές αυτές ε, οι μεγάλες επιχειρήσεις ε, αγοράζουν υπηρεσίες από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχει μια ολόκληρη αλυσίδα αξίας, ε, παγκοσμιοποιημένη πλέον, που περιλαμβάνει και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά το γραφείο μας στην Κολομβία, ευχαριστώ που με ρωτήσατε. Ναι, το ανοίξαμε και λειτουργεί απλά δεν έχει ακόμα εγγενιαστεί επισήμως. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας Επενδύσεων θέλει να έρθει στην Ποκοτά να το εγγενιάσει το γραφείο μας ο ίδιος και έχουμε δυσκολία να βρούμε την κατάλληλη χρονική στιγμή και εξαιτία ε, των εκλογών ε, δεν βρίσκαμε την κατάλληλη ημερομηνία. Πριν το τέλος του χρόνου θα είναι εγγενιαστεί. Πάντως το γραφείο μας υπάρχει και λειτουργεί και μάλιστα εντός ε, του κτηρίου της ε, αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Μας ε, ε, στήριξε η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και επίσης από την Κολομβιανή Κυβέρνηση. Ακόμα απλώ δεν, δεν έχουν γίνει επίσημα τα εγγένεια. Σε ό,τι αφορά την Κίνα είναι πολύ ευαίσθητο το ζήτημα. Μπορώ να σας να αναφερθώ σε τρεις πτυχές. γιατί κινέζικες ε, εταιρείε, ή ε, επενδυτικοί φορείς έχουν πλεονέκτημα. Πρώτον διότι έχουν ένα μακροχρόνιο, μακρόπνο όραμα, το οποίο δεν έχουμε πάντα εμείς. Εμείς ε, εξετάζουμε τις εντολές που μας έχουν δοθεί. Εγώ πολύ συχνά χρηματοδοτώ σχέδια που διαρκούν 25 χρόνια. Για τους Ευρωπαίους είναι δύσκολο να αντιληφθούν ότι ορισμένες από τις επενδύσεις, ορισμένες από τις αλλαγές που θέλουμε να προκαλέσουμε μέσω των επενδύσεων χρειάζονται χρηματοδότηση που θα πληρωθεί από αυτή αλλά και από την επόμενη γενιά. Γιατί και η επόμενη γενιά θα ζήσει τα ωφέλη. Οπότε το θέμα της αλληλουχίας ε, το έχουν πολύ καλύτερα οι Κινέζοι. Ε, δεύτερον, η προσέγγιση των Κινέζων είναι πολύ πιο κέντροσχεδιασμένη από τη δική μας ε, εστιάζουν πάρα πολύ περισσότερο και όλες τους τις δυνάμεις τις συγκεντρώνουν σε ένα συγκεκριμένο στόχο ενώ οι δικές μας δυνάμεις πολύ συχνά κατακαιρματίζονται. Τρίτον, έχουν διαφορετικούς κανόνες στους οποίους πακούν. Διαφάνεια, ας πούμε, <laughs> έχουμε πολύ διαφορετική ερμηνεία της λέξης διαφάνεια. Επίση, εμείς είμαστε τελείως ε, ανοιχτοί ε, και ζητάμε να είναι ανοιχτοί όλοι οι διαγωνισμοί προμηθειών. Ε, αυτοί έρχονται και κάνουν προσφορές για τους εργαζόμενους, για τα, τη χρηματοδότηση, όλα μαζί ένα πακέτο και εγώ ρωτάω τους υπεύθυνους εκείνες τις χώρες, είστε σίγουροι ότι παίρνετε πίσω την αξία αυτού που δίνετε. Για παράδειγμα, οι Κινέζοι χρηματοδοτούν λιμάνια σε, μια, σε ένα αριθμό χωρών ε, και αυτές οι χώρες συχνά ε, δεν μπορούν να, να, τα πληρώσουν και να τα λειτουργήσουν μετά. Οπότε τα εκχωρούν στους Κινέζους τελικά και περνάνε σε κινέζικα χέρια. Αυτή είναι η λόγια του οποίου οι Κινέζοι έχουν ένα πλεονέκτημα Βέβαια, σε ορισμένε χώρε και κυρίω στην Αφρική προ το παρόν, αντιλαμβάνονται οι υπεύθυνοι ότι δεν είναι ακριβώ προ συμφέρον του αυτό ο εναγκαλισμό, δεν θα είναι προ συμφέρον των επόμενων γενιών. Ε, αλλά πάντω σίγουρα είναι διαφορετική η προσέγγιση των Κινέζων. Σα ευχαριστούμε. Θα επανέλθουμε σίγουρα σε αυτό το σημείο. Ο κύριο Γιώργιντσεν, το λόγο. Ε, ευχαριστώ να απαντήσω σε ερωτήσεις με τη σειρά που υπευλήθησαν. Πρώτη ερώτηση. Υπάρχουν προϋποθε... μάλλον συνθήκες εργασίας στο Εκουαδόρ, στις φυτίες μπανάνας που νομιάζουν με συνθήκες δουλείας και χθε άκουσα την ερώτηση αυτή σε μια αντιπροσωπεία και όντως αυτό, αυτή την καταγγελία πρέπει να αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ σοβαρά, αλλά δεν θα πρέπει και να την καρδία κανείς να κάνει τέτοιες δηλώσεις. Στις συναντήσεις που είχαμε πέρυσι, στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, δεν είχε τεθεί ποτέ ένα τέτοιο ζήτημα. Καταγράφουμε πάντως την ανησυχία αυτή και αυτό το οποίο θα έλεγα είναι να εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν στο πλαίσιο της συμφωνίας, για, όσον για όσους κάνουν τις καταγγελίες αυτές δηλαδή, προκειμένου να επιληφθούμε του ζητήματος αυτού εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έπειτα και στα πλαίσια της συμβουλευτική ομάδας της κοινωνίας των πολιτών με την Κολομβία, το Περού και τον Ισημερινό. Και να θίξουμε το ζήτημα αυτό στην επόμενη συνάντηση που θα έχουμε μαζί τους τον Νοέμβριο. Δεύτερη τώρα ερώτηση από την κυρία Πινιέρο όσον αφορά την εφαρμογή μάλλον την έκθεση για την εφαρμογή τη Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών. Δεύτερη φορά που υποβάλλουμε τέτοια έκθεση για την εφαρμογή και όσον αφορά τη Λατινική Αμερική, αυτό το οποίο θέλουμε είναι να έχουμε μια πιο συγκρίσιμη και σφαιρική πλέον εικόνα και περιγραφή των πραγμάτων για διάφορε πτυχέ τη εφαρμογή. Για παράδειγμα, πώ χρησιμοποιούνται τα ποσοστά όσον αφορά τι προτιμήσει, για παράδειγμα, έχουμε ένα πρόβλημα με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής που δεν έχουμε την χρήση των ποσοστώσεων αυτών των προτιμησιακών. Επίσης θέλουμε να τυποποιήσουμε κάπως τα δεδομένα χρησιμοποιώντας μόνο δεδομένα της Eurostat για όλες τις χώρες και θέλουμε να διασφαλίσουμε επίσης ότι υπάρχει μια ισχυρή και αρκετά ευρεία υποβολή δεδομένων για συμφωνίες όπως αυτή με τη Χιλή για παράδειγμα ή το Μεξικό για την οποία δεν υπάρχει ρητή και επίσημη υποχρέωση υποβολής έκθεσης. Άρα και οι δύο αυτές χώρες θα συμπεριληφθούν στα δεδομένα που θα περιέχει η επόμενη έκθεσή μας. Και θέλουμε να είμαστε όσο δυνατόν και πιο σφαιρική στην έκθεση αυτή, να καλύπτουμε όλες τις πτυχές και θέλουμε να καλύψουμε κατά αυτόν τον τρόπο και την βιώσιμη ανάπτυξη όπως προβλέπει άλλωστε και ο κανονισμός για την εφαρμογή αυτών των συμφωνιών. Τώρα, να απαντήσω στην ερώτηση της κυρίας Βαν Γκράτστεν Χάιντς, η οποία είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πιο ισχυρή εφαρμογή του κλάδου εκείνου που έχει να κάνει με την βιώσιμη ανάπτυξη. Κοιτάξτε, εμεί γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή δύο πράγματα. Πρώτον, προφανώ ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα, να επενδύσουμε περισσότερου πόρου και αυτό θα το κάνουμε. δεν θα ασχοληθούμε απλώς μόνο με κάποια ζητήματα που έχουν προκύψει, αλλά θα διοργανώσουμε και περισσότερες εκδηλώσεις στις χώρες αυτές. Θα ενισχύσουμε επίσης τις δυνατότητες συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στον διαρθρωμένο αυτόν διάλογο που έχουμε. Και ξέρω ότι εσείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιμένετε από εμά να λάβουμε πιο έντονη δράση. Και έτσι λοιπόν αυτό το σχέδιο με τα 15 σημεία, το οποίο εγκρίθηκε ε, τουλάχιστον ε, επί της αρχής ότι θα πρέπει να ενσωματωθεί δηλαδή συμφωνίες αυτές, θα πρέπει να δούμε και αυτό πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Κάναμε μια συνεδρία στην προηγούμενη εβδομάδα με τις χώρες της ε, Κεντρικής Αμερικής και συμφωνήσαμε με τους εκπροσώπους της χώρας αυτής ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε ένα συγκεκριμένο, σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης. Και Κάτι αντίστοιχο θέλουμε να κάνουμε και με τον Σημερινό και με την Κολομβία στην συνεδρίαση που θα έχουμε τον Νοέμβριο. Ένα από τα ζητήματα που θα θίξουμε είναι η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στο Περού. Γιατί όπως ακούσαμε το Περού δεν τηρεί τις δεσμεύσεις του σε σχέση με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Και οι συμφωνίε αυτέ, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, μα δίνει όντω τη δυνατότητα να προωθήσουμε περισσότερο την ε, συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών και να ασχοληθούμε και εμεί περισσότερο με αυτό το ζήτημα για πιο σοβαρά. Τώρα, αν υπάρχουν κατευθυντήριε γραμμέ όσον αφορά τι αντιπροσωπείε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε ότι ε, έχουμε προφανώ συγκεκριμένε κατευθυντήριε γραμμέ για την αντιπροσωπή ουσιαστικά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τη ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση. Τα όσα έχουμε πετύχει αυτή τη στιγμή στην Κολομβία έχουν να κάνουν με την έμφαση που εμείς δώσαμε ως αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί για το πώς θα πρέπει να εφαρμοστούν αυτές οι συμφωνίες. Έχουμε εξαιρετική σχέση με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει να κάνει μόνο με την πολιτική και το εμπόριο. Πολλέ φορέ το εξετάζουμε στα επιμέρου του στοιχεία, όντω βιώσιμη ανάπτυξη όσον αφορά το εμπόριο, όσον αφορά τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Άλλε φορέ όμω υπάρχουν ξεχωριστέ πρωτοβουλίε για την ειρηνευτική διαδικασία, για παράδειγμα. Στην Κολομβία, για παράδειγμα, έχουμε μια εμπορική συμφωνία για την ειρηνευτική διαδικασία. Δηλαδή προσπαθούμε να δούμε πώς η εμπορική αυτή συμφωνία μπορεί να συμβάλλει και να προωθήσει την ειρηνευτική συμφωνία. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δώσετε να συμμετάσχω σε αυτή τη συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ πολύ και με πείσετε ότι ζούμε σε ένα τέλειο κόσμο ευχαριστήσω όλους τους uh, συμμετέχοντες και στα δύο πάνελ. Πολύ έντονη συζήτηση που έγινε, πολύ ενδιαφέρουσα επίσης. Ζήτησε κάποιος να κάνει μία ακόμα παρατήρηση, σύντομα. Αν μου επιτρέπετε, είμαι ο πρέσβης του Περού. Αν μπορούσα να έχω ένα λεπτό για να σχολιάσω δύο-τρία θέματα σχετικά με ορισμένα πόσα ελέγχθησαν σε σχέση με ένα από τα προβλήματα της χώρας μου. Πιο συγκεκριμένα για τα DAG, τα, τις ομάδες ε, συμβουλευτικές, ε, εθνικές συμβουλευτικές ομάδες. Σύμφωνα με το άρθρο 281 της ε, Συνθήκης Ελεύθερων Συναλλαγών που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε μέρος θα διαβουλεύεται με τις εθνικές ομάδες ή επιτροπές που σε εργασιακά περιβαλλοντικά θέματα ή θέματα βιώσιμης ανάπτυξης ε, διαθέτουν στη χώρα τους. Και όταν δεν υπάρχουν τέτοιου είδους ομάδες θα δημιουργούνται όλα αυτά σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της κάθε χώρας. Στο Περού υπάρχουν διάφορες ομάδες ε, που συνδέονται με αυτά τα θέματα. Εθνικό Συμβούλιο Εργασίας, ε, Εθνικό Συμβούλιο ε, Ασφάλειας στο χώρο ένα Συμβούλιο Βιολογικής Ποικιλότητας, Βιοποικιλότητας. το σε ορισμένες φορές απλώς ε, επικεφαλής τίθεται το κράτος. Ε, ε είπε ο Ιταλός συνάδελφος. Ε, να σας πω όμως ότι πριν από μερικές εβδομάδες οι αρχές του Περού και πιο συγκεκριμένα το Υπουργείο Εργασίας υπέβαλαν πρόταση έτσι ώστε το Εθνικό Συμβούλιο εργασίας ε, που είναι αυτό που ε, έχει ε, τη μεγαλύτερη ποικιλία οργανώσεων στο εσωτερικό του να προεδρεύεται, να έχει επικεφαλή σε άτομο το οποίο θα είναι αυτόνομο από τον κρατικό μηχανισμό. Εμείς δεν ερμηνεύουμε το άρθρο 281 ως να, ότι μας υποχρεώνει να δημιουργήσουμε ε, μία ο εσωτερική συμβουλευτική ομάδα ε, ίδια με ε, αυτήν που έχουν δημιουργήσει άλλα μέρη της συμφωνίας. Κάθε χώρα που έχει υπογράψει συμφώνιας σύμφωνα με τη δική της εσωτερική νομοθεσία, θα πρέπει να ιδρύει τις ομάδες DAG. Άλλο ένα σχόλιο. Γι' αυτό το λόγο ε, έχει υποβληθεί μια, ε, ένα παράπονο, μια καταγγελία από μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, καταγγελία την οποία εξετάζει τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το κράτος. Αυτό είναι απόδειξη ότι οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα έχουν δικαίωμα να εκφράζουν την άποψή τους και να χρησιμοποιούν τους όρους της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών. Ευχαριστώ. Ε, Η ακρόαση αυτή δεν αφορά το Περού βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, έχουμε το επόμενο θέμα το οποίο αφορά την έκθεση εφαρμογής για την Κολομβία και το Περού. Εκεί θα συζητήσουμε και το Περού πιο συγκεκριμένα. Το συζήτησα και με τον Υπουργό Εμπορίου σας. Έχουμε διαφορετικές απόψεις, αποκλείουν σας απόψεις, αλλά εν πάση περιπτώσει ο διάλογος είναι καλός. Ευχαριστούμε πολύ για τους συμμετέχοντες στο πάνελ. Χρήσιμα τα όσα μας είπαν και σίγουρα θα επανέλθουμε στο ζήτημα. Το Η εφαρμογή της ε, συμφωνίας για την Κολομβία και το Περού που υπεγράφει πριν από πέντε χρόνια. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Φίσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με την Κολομβία και το Περού έχει εφαρμοστεί προσωρινά για πέντε χρόνια. Οπότε καλή στιγμή για να κάνουμε μια αξιολόγηση της εφαρμογής αυτής. Υπεγράφει στις 26 Ιουνίου του 12 και άρχισε να ισχύει προσωρινά με το Περού από τον Μάρτιο του 13 και με την Κολομβία από τον Αύγουστο του 13 και έδωσε τη σύμφωνη γνώμη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την σύναψη αυτής της συμφωνίας στις 11 12 του 2012 και τον Ιανουάριο του 2017 συμπεριλήφθηκε ο Ισημερινός αυτή τη συμφωνία. Κάτι που έχει να κάνει με τη στρατηγική και εμπορική σημασία. Είναι προτεραιότητα η εξέταση των συμφωνίων αυτών για την Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο. Πρέπει να τις ε, παρακολουθούμε, όχι μόνο κατά τη διαπραγμάτευση, αλλά και κατά την εφαρμογή. Χθες, όπως υπόθηκε, είχαμε μια συνάντηση της ομάδας ε, επίβλεψης με τις ε, χώρες ε, των Άνδεων όπου συμμετείχαν και εκπρόσωποι από την καλλιέργεια μπανάνας και συλλέγουμε και στοιχεία επιτόπου. Μία αντιπροσωπεία της ΣΥΝΤΑ πήγε το Φεβρουάριο 12 με 16 στην ε, Κολομβία και το Περού και τα αποτελέσματα θα τα δείτε στην έκθεση για την εφαρμογή και την περασμένη Δευτέρα η Γραμματεία μοίρασε την επίσημη έκθεση τη Επιτροπή. Δυστυχώ δεν μπόρεσα να συμμετάσχω σε αυτή την αποστολή γιατί χρειάστηκε να κάνω μια εγχείρηση. Σήμερα η Επιτροπή μας εξετάζει την έκθεση εφαρμογής της ε, συμφωνίας με την Κολομβία και τον Περού. Θα σας παρουσιάσω τις γενικές μου ιδέες για την έκθεση που θα παρουσιάσω στην επόμενη συνεδρίαση στις 27 Σεπτεμβρίου και θα την ψηφίσουμε στην Ίντα τον Νοέμβριο. Αγαπητοί συνάδελφοι, θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Όπως είπε και ο πρόεδρός μας, μισογεμάτο το ποτήρι. Δεν έχει αυξηθεί βέβαια το διμερές εμπόριο, αλλά η συμφωνία εν μέρη αντιστάθμισε τις αρνητικές τάσεις του διεθνούς εμπορίου, συνέβαλε στην ε, οικονομική σταθερότητα, τον εξυγχρονισμό και τη διαφοροποίηση των εξαγωγών στην Κολομβία και τον Περού. Οι εμπορικέ και επενδυτικέ ροέ, γενικά είναι θετικέ. και αμοιβαία επωφελεί. Τονίζω ότι οι εξαγωγέ γεωργικών προϊόντων της Ένωσης αυξήθηκαν ουσιοδό και προ τι δύο χώρες. Η εφαρμογή της συμφωνία είναι σημαντικό εργαλείο για να βελτιωθεί η πρόσβαση για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε αυτές τις αγορές. Όχι μόνο η καταργή τους ε, δασμούς, αλλά καταργεί και τις, ε, τους άλλους εμπορικούς φραγμούς. Η Επιτροπή μας έδωσε λεπτομεριακά στοιχεία για το εμπόριο και τις επενδύσεις και ελπίζω να λάβουμε πληροφορίες και για την επίπτωση της συμφωνίας στις μικρομεσαίες. Η ετήσια έκθεση εφαρμογής της Επιτροπής μας δίνει τη δυνατότητα να θεωρήσουμε ότι είχε πολύ θετικέ εξελίξεις για τις μικρομεσαίες στις δύο αυτές χώρες, για την Κολομβία 2.002 εταιρείες εξήγαγαν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016 ενώ ήταν ε, γύρω στις 1.500 το 2011. Από τότε που ε, άρχισε να λειτουργεί αυτή η συμφωνία 2.200 και ε, επιχειρήσεις παραπάνω από τις χώρες αυτές ή μάλλον συγκεκριμένα από το Περού εξήγαγαν προς την Ένωση. Βέβαια υπάρχουν ακόμη ορισμένα προβλήματα σε εμπορικές σχέσεις. Θα τα αναφέρουμε στην έκθεση και πρέπει να τα υπερβούμε σύντομα. Γιατί αντιβαίνουν στη συμφωνία. Για παράδειγμα, προστατεύονται κάποιες ε, γεωγραφικές ενδείξεις. Ο διάλογος για το εμπόριο και, το βιώσιμο, και τη βιώσιμη ανάπτυξη με τους εταίρους μας και με την ε, κοινωνία των πολιτών έχει αυξηθεί. Είναι σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εφαρμόζεται η διεθνή εργασιακή και περιβαλλοντική νομοθεσία. Θεωρούμε ότι οι εμπορικές αυτές συμφωνίες μας βοηθούν και πολιτικά να βελτιώσουμε την κατάσταση στις χώρες αυτές. Αλλά παράλληλα, τα μέτρα για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι σημαντικό για να προστατεύσουν τις ε, δικές μας επιχειρήσεις από το κοινωνικό και περιβαλλοντικό dumping που μπορεί να κάνουν κάποιες εταιρείε εκεί. Ζητάμε προγράμματα δράσης από τις χώρες αυτές για να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη. Είχαμε ζητήσει τότε, πριν εγκρίνουμε τις συμφωνίες. Και οι δύο χώρες υπέβαλαν αυτά τα προγράμματα δράσης. Αυτό εκφράζει την καλή τους θέληση για τους τομείς αυτούς. Τονίζω επίσης ότι είναι οι μόνες χώρες από τις οποίες απέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έναν οδικό χάρτη πριν εγκρίνει τι συμφωνίε. Μέσω τη έκθεση θα εξετάσουμε πώ έχουν εφαρμοστεί αυτά τα προγράμματα δράση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θεωρώ ότι και η Κολομβία και το Περού σημειώνουν ουσιώδη πρόοδο και αν δεν είχε υπάρξει αυτή η συμφωνία δεν θα είχαν υπάρξει τόσε πρόοδοι. Να μην ξεχνάμε όμω ότι πολλά ακόμη πρέπει να γίνουν για θέματα όπω η καταπολέμηση τη διαφθορά, η προστασία του περιβάλλοντο, καλύτερα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, συνδικαλιστικές ελευθερίες, επιθεώρηση εργασίας και οι άτυπες μορφές εργασίας. Στο Περού η άτυπη εργασία είναι 73% και στην Κολομβία 58% και επίσης η παιδική εργασία. Όμως και οι δύο χώρες πέρασαν από πολύ δύσκολες περιστάσεις. Αν εφαρμόσουμε ευρωπαϊκές προδιαγραφές βέβαια δεν είναι ιδανική η κατάσταση. Αλλά Πρέπει να ενθαρρύνουμε αυτέ τι φιλικέ χώρε για να συνεχίσουν να εργάζονται προ τη σωστή κατεύθυνση και να ξέρουν ότι μπορούν να βασίζονται και στη δική μα βοήθεια. Άλλο σημαντικό στοιχείο, ήδη αναφέρθηκε για μα, είναι η δημιουργία αυτών των εσωτερικών συμβουλευτικών ομάδων που να είναι πραγματικά ανεξάρτητε για να παρακολουθούν την εφαρμογή των συμφωνιών και να προωθούν το διάλογο. Συγχαίρω την Κολομβία για την απόφαση να δημιουργήσει αυτήν την ε, ομάδα που είναι ανεξάρτητη από την κυβέρνηση και για το διορισμό 908 επιπλέον επιθεωρητών. Και καλό το Περού να κάνει κάτι παρόμοιο. Ακούσαμε και τον πρέσβη. Ότι είναι ακριβώς ε, σε φάση δημιουργίας αυτών των θεσμών. Είναι σημαντικό το ότι μπήκε η Κολομβία στις 30 Μαΐου στον ΟΣΑ ο οποίος είναι την Κολομβία για τις εντυπωσιακέ μεταρρυθμίσεις, για παράδειγμα, στο δικαστικό σύστημα για τη μείωση των ατύπων μορφών εργασίας. Η Κολομβία, η Κολομβία έκανε σημαντικό βήμα για να λειτουργούν καλύτερα οι ε, κρατικές επιχειρήσεις και για να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα διαφθοράς και δωροδοκίας. Αυτά, συνάδελφοι, και με βάση και τις παρατηρήσεις σας και τη βοήθεια όλων των σκιωδών θα αρχίσω να εργάζομαι για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Καλώς ορίζω τον πρέσβη του Περού και τους εκπροσώπους της πρεσβείας της Κολομβίας. Ε, με ικανοποίησε η παρουσίαση της έκθεσης εφαρμογής του κρυοφύσας. Μόλις ε, πάρουμε το έγγραφο στα χέρια μας θα δούμε αν χρειάζεται να υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες. Πάντως είναι προς σωστή κατεύθυνση κινείται. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε αφενός ε, τα ωφέλη που προέκυψαν από τη συμφωνία με το Περού και την ε, Κολομβία. Πώς, τι ακριβώς βελτιώθηκε και πώς ακριβώς εφαρμόστηκαν αυτές οι συμφωνίες. Και από την άλλη μεριά να εντοπίσουμε τις ε, αδυναμίες που απομένουν και που πρέπει να διορθωθούν. Έχω πει και στο παρελθόν το εξή. Και στη Συμφωνία του Περού και στη Συμφωνία της Κολομβίας καλό είναι να συμπεριλάβουμε και εργαλεία τα οποία ήδη υπάρχουν Συμφωνία με το Μεξικό. Προκειμένου να διευκολύνουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να τις ενημερώνουμε μέσω, για παράδειγμα, ενιαίων θηρίδων και με άλλα εργαλεία τα οποία διαθέτουμε ήδη στη συμφωνία με το Μεξικό. Πρέπει να διαδώσουμε περισσότερο την πληροφορία και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αυτές του Περού και της Κολομβίας με ανησυχεί λίγο το εξής. Η... Θα πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή της συγκοινωνίας των πολιτών. Ο κ. Γιολιάνο είπε κάτι προηγουμένως με το οποίο συμφωνώ. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο διάλογος με την κοινωνία των πολιτών είναι κάτι θετικό που προκύπτει από τις συμφωνίες. Δηλαδή οι εμπορικές συμφωνίες έχουν ως σκοπό να βελτιωθεί η ζωή των εργαζομένων, ε, οι εργασιακές τους συνθήκες και η ανταγωνιστικότητά τους. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να οι βασικοί φορείς να ενημερώνονται και να τους δίνεται ευκαιρία να συμμετέχουν. Οπότε περιμένουμε το κείμενο του κ. Φίσας και θα συνεργαστούμε μαζί του. Thank you, Mr. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ και εγώ να συμμετέχω στην συζήτηση αυτή για την πρώτη έκθεση εφαρμογής και εγώ έχω ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό εδώ και πολύ καιρό και μάλιστα Ήμουν εδώ όταν πρωτοσυστάθηκαν οι συμφωνίες αυτές, όταν τις θεσπίσαμε για πρώτη φορά. Χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν που υπάρχουν και που εφαρμόζονται και που έχουμε φτάσει στο σημείο που μπορούμε να αξιολογήσουμε τα πρώτα έμπρακτα αποτελέσματα αυτών των συμφωνιών. Τώρα, όσον αφορά την Κολομβία, εμπορικές επιπτώσεις. Αν συγκρίνουμε τα δεδομένα που έχουμε με τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Νοτιού Κορέα θα μπορούσαμε ίσως να τα είχαμε πάει κάπω καλύτερα. Διότι η συμφωνία αυτή που ανέφερα τώρα με την Νότια Κορέα σημείωσε άμεση επιτυχία, ενώ εδώ τώρα με την Κολομβία βλέπουμε ότι υπάρχει μια κάποια καθυστέρηση στα θετικά αποτελέσματα, μόλον ότι το δυναμικό εδώ πέρα είναι τεράστιο λόγω του πλούτου που έχει η Κολομβία και λόγω των, του μεγέθους της και έχει επίση ένα πολύ νέο εργατικό δυναμικό. Βλέπουμε όμως ότι έχουν ήδη διαφοροποιηθεί πάρα πολλοί εξαγωγές της Κολομβίας. Αυτό είναι πολύ θετικό, βρίσκεται σε θετικό δρόμο. Αναφερόμαστε εδώ πέρα όχι μόνο σε καύσιμα και σε άλλες πρώτες και μεταλλεύματα, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν και γεωργικά προϊόντα. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συμφωνία αυτή, μάλλον να προβάλλουμε τη συμφωνία αυτή και στις δύο πλευρές και να δείξουμε σε επιχειρήσεις και δύο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πώς μπορούν να αποφεληθούν από τη συμφωνία αυτή. Γιατί δεν νομίζω ότι αυτό έχει γίνει ακριβώς ακόμα πλήρως. Και υπάρχουν και κάποιες συγκεκριμένε δυσκολίες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. δυσκολίες μη δασμολογικής φύσης για παράδειγμα το ότι είναι υπερβολική η φορολόγηση όσον αφορά τα υνοπνευματώδη ποτά και επίσης δεν είναι πολύ εύκολο για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς κρατικών προμηθειών. Όσον αφορά τώρα τη συμφωνία με το Περού, Εκεί έχουμε πάλι κάποια ανάμεικτα αποτελέσματα, τουλάχιστον στην αρχή και μάλιστα στην πολύ πολύ αρχή τα πρώτα χρόνια μειώθηκαν τα ποσοστά του εμπορίου. Τώρα βλέπουμε ότι τα πράγματα πηγαίνουν κάπως καλύτερα, έχει αυξηθεί το εμπόριο κατά τη διάρκεια του 2017, έχουμε διαφοροποίηση των εξαγωγών της χώρας αυτής και έχουν αυξηθεί επίσης τα προϊόντα αυτά τα οποία φέρουν μεγαλύτερη πλέον προστιθέμενη αξία. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι ανάμεσα στις δύο χώρες το Περού είναι αυτό το οποίο έχει αποκομίσει τα περισσότερα ωφέλη, καθότι έχει μάλιστα και πλεονέκτημα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώ όμω πάλι υπάρχουν επιχειρήσει οι οποίε δεν γνωρίζουν πολύ καλά τι θετικέ πτυχέ αυτή τη συμφωνία. Θα πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο και τι επιχειρήσει, κυρίω από την ευρωπαϊκή πλευρά, για τη συμφωνία αυτή. Αυτά είχα να πω εν συντομία και προσβλέπω στο σχέδιο έκθεση που θα υποβάλει ο εισηγητή και προφανώ θα συνεργαστώ και μαζί του και με του υπόλοιπου σκιώδει εισηγητέ για να βρεθεί μια θετική έκθεση η οποία θα είναι αμοιβαία αποδεκτή. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Σόλτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με του προλαλήσαντε και εγώ. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα ήθελα να διαβάσω το σχέδιο έκθεσης που θα υποβάλει ο εισηγητής και αυτό διότι πιστεύω ότι οι δύο αυτές συμφωνίες μας έχουν απασχολήσει πάρα πολύ καιρό εδώ πέρα στο πλαίσιο της Επιτροπής. Ξέρετε ότι κάναμε πάρα πολλές ανταλλαγές απόψεων για τις εμπορικές πτυχές αλλά και τις πολιτικές πτυχές των δύο αυτών συμφωνιών. θυμάστε κάποιες από τις αρχικές προκλήσεις που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε και τα διδάγματα που μπορέσαμε να αντλήσουμε από την επίσκεψη στην Κολομβία και το Περού. Αν θέλετε, η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις εμπορικές αυτές πτυχές της συμφωνίας με την ειρηνευτική διαδικασία είναι πολύ σημαντική. Αυτό το είπαν όλοι. Υπάρχει μια έντονη διασύνδεση ανάμεσα αυτές τις δύο πτυχές. και νομίζω ότι η πτυχή αυτή θα πρέπει να συμπεριληφθεί από τον εισηγητή στο σχέδιο έκθεσης. Και ξέρετε ότι ε, η κοινωνία ήταν εντελώς διχασμένη. Το ότι έχουμε ουσιαστικά αυτούς οι οποίοι ζουν σε πόλεις, στα μεγάλα αστικά κέντρα ή στην πρωτεύουσα και όλους αυτούς οι οποίοι κατοικούν στην Ήπεθρο. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ε, εντελώς διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά την εμπορική αυτή συμφωνία. Οι απόψεις τους αποκλίνουν πάρα πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι δεν έχουν δει ακόμα τα ωφέλη από την αγροτική μεταρρύθμιση. Και υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι δεν έχουν επωφεληθεί καθόλου από τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στο παραγωγικό μοντέλο της Κολομβίας. Έτσι λοιπόν, όταν καλούμεθα να αποτιμήσουμε τα τελευταία αυτά πέντε χρόνια, Μάλλον θα πρέπει επίσης ε, να δούμε πώς θα συνεχιστεί η εφαρμογή της συμφωνίας αυτής στο μέλλον, προς όφελος όμως ε, όλων για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη όλων των πολιτών. Γιατί κάθε πολίτης ε, αποτιμά ουσιαστικά την αξία των συμφωνιών αυτών σε προσωπικό επίπεδο και γενικό επίπεδο και θα πρέπει ουσιαστικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση να φαίνεται ότι είναι ένας θεμητό σωστό εταίρος με την Κολομβία και το Περού. Πρώτον αυτό. Ας ασχοληθούμε έπειτα το εργασιακό κεφάλαιο και να δούμε λίγο και τον άτυπο τομέα εργασίας όπου εδώ πέρα δεν έχουμε τις αναμενόμενες βελτιώσεις. Δεν έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι θα ήταν ε, ιδιαίτερα χρήσιμο οι διάφορες πρεσβείες να μας δίνουν πλέον μόνιμες σταθερές πληροφορίες ε, όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Είπατε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να εμπλέξουμε περισσότερο την Κολομβία στο κεφάλαιο αυτό που έχει να κάνει με το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ενδεχομένως λοιπόν θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε και κάποιες τέτοιες ιδέες και σκέψεις σε αυτό το σχέδιο έκθεσης. Όσον αφορά την δική μου πολιτική ομάδα, πρέπει να σας πω ότι προφανώς ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ να συνεργαστούμε με τον εισηγήτη και τους κοιόδης εισηγητές και να καταφέρουμε έτσι από κοινού να βελτιώσουμε την έκθεση αυτή και να δούμε τελικά ποια είναι τα θετικά στοιχεία ή που πρέπει να κάνουμε κάποιες τροποποίησεις ή ενδεχομένως κάποια προβλήματα να τα έχουμε ήδη επιλύσει. Αυτά είχα να πω επί του παρόντος. Εγώ πραγματικά είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο μετά από αυτά που είπατε ότι δηλαδή καλύψατε στην έκθεσή σας όλες αυτές τις πτυχές που συζητήσαμε εδώ τα τελευταία χρόνια στην Επιτροπή μας. Θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται όλες αυτές στην τελική έκθεση σίγουρα. Και πρέπει να πω ότι ε, η Επιτροπή μας θα πρέπει να καταφέρει να γίνει μόνιμος παρατηρητής της εφαρμογής των δύο αυτών συμφωνιών. Δηλαδή να μην ασχολούμεθα με τις συμφωνίες αυτές μόνο κάθε πέντε χρόνια, αλλά να έχουμε ένα πιο μόνιμο μηχανισμό, μια πιο μόνιμη διαδικασία παρακολούθηση τη εφαρμογή των δύο αυτών εμπορικών συμφωνιών. Να έχουμε άμεση ανταλλαγή απόψεων, για παράδειγμα, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την DigiTrade, με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Και να βλέπουμε έτσι σε συστηματική συνεχή βάση που υπάρχουν περιθώρια βελτίωση για αυτέ τι συμφωνίε. Thanks a lot. This was a very... Πολύ ευγενική η συζήτηση. Ε, δεν είναι πάντα έτσι, αλλά γενικά είμαστε πολύ ευγενεί ο ένας σχέση με τον άλλο. Κύριε Γιώργενσεν. Thank you uh, uh. από πλευράς μου. Συμφωνώ με τον κύριο Φίσας που λέει ότι το ποτήρι είναι μισογεμάτο. Πολλά έχουμε κάνει και πολλά απομένουν. Σίγουρα δεν μπορούμε να επαναπαυθούμε. Ούτε εμείς ούτε η άλλη πλευρά. Η συμφωνία αυτή μπορεί να προχωρήσει μόνο αν και οι δύο πλευρές το επιθυμούν και επενδύσουν προσπάθειες αυτό. Αν δούμε λίγο τα νούμερα. Από, σε μια πρώτη ανάγνωση, κανείς μπορεί να πει ότι ε, το εμπόριο δεν έχει αυξηθεί τόσο πολύ όσο, με, όσο σε άλλες συμφωνίες, ε, αλλά αν το δούμε πιο βαθιά, τα αγροτικά προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κολομβία αυξήθηκαν κατά 95% από το 2011 2017. Ε, το ίδιο και οι εξαγωγές στο Περού αυξήθηκαν κατά 75% στην ίδια περίοδο. Μόνο πέρσι ε, ε, ε, αυξήθηκαν και οι εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το νησιμερινό. Και οι εξαγωγές πρώτων υλών από αυτές τις χώρες βέβαια μειώθηκαν, αυξήθηκαν, συγγνώμη, και η Κολομβία αύξησε τα, τις εξαγωγές τροφίμων κατά 50-45%, το Περού κατά 35%, Οπότε αυτές οι χώρες γίνονται όλο και λιγότερο ε, εξαρτώμενες από, την, από το εμπόριο πρώτων υλών. Εξάγουν πλέον και άλλου είδους προϊόντα. Έχουμε ένα θέμα πρόσβασης αγορές, το οποίο το λύσαμε. Με την Κολομβία είχαμε ένα θέμα πρόσβαση στι ε, κρατικές προμήθειε σε, σε περιφερειακό επίπεδο. Είχαμε ένα θέμα με τα αλκοολούχα ποτά. Ε, ε, η Κολομβία επίσης ακύρωσε προτιμησιακή πολιτική που είχε ενώ το Περού Έλυσε επίσης διάφορα προβλήματα σε σχέση με, τις, με προτιμησιακό καθεστώς, με δασμούς που ε, παρέμεναν κλπ. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν εκκρεμή θέματα. Για παράδειγμα, το Περού και η, το Εκουαδόρ και το Ισημερινός ε, ε, σε σχέση με τις μεταφορές κατάργηση ενός ε, νόμου που ε, ευνοεί τις εθνικές ε, εταιρείες κλπ. Η βιώσιμη ανάπτυξη επίσης θα είναι κάτι στο οποίο θα εστιάσουμε στα επόμενα χρόνια. Ήδη στην Κολομβία στάθηκαν οι εσωτερικές συμβουλευτικές ομάδες και με το Περού περιμένουμε παρόμοιες, ε, παρόμοια πρόοδο έτσι ώστε να λειτουργήσουν σωστά οι μηχανισμοί διαβούλευσης. Ε, Ο σημερινός τώρα βέβαια ξεκινάει, αλλά η Κολομβία έχει βελτιώσει πολύ την θέση της και πρέπει να δούμε αν αυτές οι ομάδες πραγματικά δίνουν αποτελέσματα επί της ουσίας. Εμείς πάντως προσεγγίζουμε το θέμα με τρόπο συνενετικό, σαν να είμαστε στο ίδιο τρένο και οι δύο πρέπει να δουλέψουμε προς την ίδια κατεύθυνση για να προχωρήσει το τρένο αυτό. Και μόνο έτσι θα πετύχουμε. Λοιπόν, εκπρόσωπος ε, της ε, πρεσβείας της Κολομβίας, η κυρία Αντριάννα Βάργας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε ένα κόσμο όπου η σύγκρουση μεταξύ κοινωνιών είναι κάτι συνηθισμένο, ε, είναι σημαντικό ότι η Κολομβία κατάφερε να ολοκληρώσει τη διαδικασία του πολέμου που κράτησε 50 χρόνια με 8 εκατομμύρια θύματα και 250.000 νεκρούς. Όχι μόνο σταμάτησε η σύραξη, αλλά ξεκίνησαν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για να ε, εκριζωθούν τα αίτια της βίας, όπως η ανάπτυξη της υπαίθρου, η συμμετοχή στην πολιτική ζωή, οι παράνομες καλλιέργειες και πρώτα απ' όλα πώς θα εγγυηθούμε τα, τα δικαιώματα των θυμάτων. Θυμίζουμε ότι τα προηγούμενα μέτρα είχαν εδαφική ε, εστίαση. Δημιουργούμε 16 ε, σχέδια ανάπτυξης στι περιοχέ που εδίχησαν περισσότερο από την ε, σύραξη, που είναι πάνω από 30% του εδάφους μας. Η επίτευξη της συμφωνίας ήταν πολύ δύσκολη, τώρα έχουμε μεγαλύτερη πρόκληση ακόμη την εφαρμογή. Δηλαδή πώς θα αρχίσουν να λειτουργούν όλα αυτά τα προγράμματα, πώς θα μπορέσουν αυτές οι περιοχές που ήταν αποκομμένες να ενταχθούν ε, στη ζωή της χώρας. Τον Αύγουστο θα έχουν κλείσει πέντε χρόνια της ε, προσωρινής εφαρμογής της Συμφωνίας ε, Ελευθέρου Εμπορίου. Έτσι ενισχύθηκαν οι δεσμοί που υπήρχαν μεταξύ χωρών που έχουν τις ίδιες δημοκρατικές αξίες, ελεύθερο εμπορίου και ε, κράτους δικαίου. Είναι λοιπόν μια μεγάλη ευκαιρία ούτω ώστε το εμπόριο να βοηθήσει την ειρήνη για να έχουμε περισσότερες επενδύσεις που θα μας βοηθήσουν να ενισχύσουμε την οικονομία και να οικοδομήσουμε την ειρήνη σε αυτές τις περιοχές. Και αντίστροφα, οι παραγωγικές δυνατότητε αυτών των περιοχών επίσης θα ενισχύσουν τις εμπορικές συναλλαγές. Αυτό το αποκαλούμε στην πρεσβεία γάμος μεταξύ της Συμφωνίας Ειρήνης και της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών. Είναι μια πραγματική ευκαιρία για να δημιουργήσουμε συνδέσεις που θα μας επιτρέψουν να κερδίσουμε όλοι. Λοιπόν, ε, αξιολογούμε πώς εφαρμόστηκε η συμφωνία μας. Θεωρούμε ότι ο απολογισμός είναι ιδιαίτερα θετικός. Το αναγνώρισε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την ε, ομιλία που έκανε ε, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Η Κολομβία η, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο δεύτερος προορισμός των εξαγωγών της Κολομβίας μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες με 14% και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επίσης ο τρίτος ε, ε, εξαγωγέας προς την Κολομβία με 15% μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. 78% των εξαγωγών φρούτων της Κολομβίας γίνεται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ωφελούνται από αυτή τη συμφωνία κατά το 2017 1.155 επιχειρήσεις μας εξήγαγαν στην Ένωση προϊόντα που δεν είναι εξόριξης και από το 1900 από αυτές κάποιες είναι μικρομεσαίες και άλλες είναι πολύ μικρές. Πέρυσι το 11,3% το 11,3% των ε, επιχειρήσεών μας εξήγαν στην Ένωση. Αλλά έχουμε ακόμη πολύ μεγαλύτερο δυναμικό. Η Συμφωνία για την Ειρήνη θα αυξήσει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητές μας. Τώρα, για την εφαρμογή της συμφωνίας έχουν υπάρξει σημαντικές ε, πρόοδοι σε κάποιες επιτροπές όπως για τα υγειονομικά και φυτοοικονομικά όπου υπήρξε μια φιλική επικοινωνία μεταξύ των υγειονομικών αρχών δημιουργήθηκε μια ενοποιημένη διαδικασία μεταξύ της ΛΥΚΑ και της Λιμπίμα για τις ε, ευρωπαϊκές εισαγωγές και για βασικά γεωργικά προϊόντα για την Ένωση. Η Κολομβία επίσης ε, τήρησε τις υποσχέσεις της μέσω αλλαγής στην νομοθεσία για να υπάρχει περισσότερη πρόσβαση στην αγορά για τα ενοπληματόδη, για τα φορτηγά και για τα πνευματικά δικαιώματα. Άλλες υποπιτροπές όμως ε, πρέπει να σημειώσουν μεγαλύτερη πρόοδο όπως η υποπιτροπή για την διευκόλυνση του εμπορίου όπου θέλουμε να υπάρξει πιο δυναμική πρόοδος και για την ε, πνευματική διοκτησία όπου προστατεύονται 117 ε, ονομασίες προέλευσης της Ένωσης από την πρώτη μέρα εφαρμογής της συμφωνίας, ενώ δεν προστατεύονται οι δικές μας ονομασίες προέλευσης. Τώρα, για να προχωρήσει η συμφωνία έχουμε δύο προκλήσεις ενώπιόν μας. Πρώτα απ' όλα ε, οι ποσοστώσεις ε, που υπόκειται σε δασμούς. Χρησιμοποιούμε κυρίως το 85% για την ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο. Επίσης, έχουμε κάποια προβλήματα πρόσβασης των δικών μας ε, αγροβιομηχανικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά. Καταλαβαίνουμε την ανάγκη που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει υγειονομικές προδιαγραφές για κάποια ευαίσθητα προϊόντα. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν σωστοί ε, κανόνες του παιχνιδιού θέλουμε να συμμορφούμεθα προς αυτές τις προδιαγραφές, αλλά χρειαζόμαστε καλύτερη κατανόηση των δυσχεριών που έχουμε για να συμμορφωθούμε και περισσότερη τεχνική βοήθεια. Το κάδμιο στο κακάο, για παράδειγμα, είναι ένα καλό παράδειγμα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η παραγωγή για την ε, κατάστασή μας τώρα, αλλά η παραγωγή μας έχουν σοβαρά προβλήματα λόγω των προδιαγραφών που θα αρχίσουν να ισχύουν από του χρόνου. Άλλο παράδειγμα. Ε, Φινικέλαιο. Ανησυχούμε ιδιαίτερα για τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό. Όπως και για το κάδμιο. Καταλαβαίνουμε την ανησυχία σας για τη βιωσιμότητα των, ε, των πόρων μας. Αλλά νομίζω ότι δεν ισχύει το επιχείρημα αυτό για την περίπτωση της Κολομβίας. Το φινικέλαιο έχει, ε, καλλιεργείται με μηδέν αποψήλωση των δασών. Το πρόβλημά μας είναι ότι έχουμε πολλές χέρσες γέες λόγω ακριβώς της ε, ένοπλης ε, που είχαμε. Το, οι φίνικες και μας επιτρέπουν να αξιοποιήσουμε αυτές τις γέες και προστατεύουν το περιβάλλον. Χάρη ε, στο πρόγραμμά μας για το, την ε, καλλιέργεια του, των φινίκων αυξάνεται και η βιοπικιλότητα στις περιοχές όπου καλλιεργούνται. Είμαστε πεπισμένοι ότι υπάρχουν λύσεις για να κερδίζουν όλοι. Και το περιβάλλον πάνω απ' όλα. Ένα λεπτό ακόμη. Βεβαίως ε, έχουμε συμμορφωθεί και με το κεφάλαιο 9 για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο στο διάλογο με την κοινωνία των πολιτών, όπω ε, αναγνώρισαν και οι προηγούμενοι ομιλητέ. Υπάρχει ένα απόλυτα ανεξάρτητο συμβουλευτικό σώμα. Τώρα δεν έχω χρόνο για να μιλήσω για ε, εργασιακά θέματα. Αλλά θέλω να τονίσω ότι για πρώτη φορά οι εργαζόμενοι στον επίσημο τομέα είναι η πλειοψηφία των εργαζόμενων στις ε, πόλεις. Έχουμε επίση πολύ περισσότερου, έχουμε διπλασιάσει του επιθεωρητέ εργασία. Και άλλη πρόοδο έχει σημειωθεί. Για το περιβάλλον, επίση έχουμε σημειώσει πρόοδου. Για την ε, προστασία των δασών, έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα ελίτ για την καταπολέμηση της αποψήλωσης και επίσης ειδικού εισαγγελεί. Και προσπαθούμε να έχουμε και αναλλακτικές χρήσει ε, χρήσεις γης αλλά πρέπει να τονίσω ότι η ένταξή μας στον ΟΣΑ είναι μεγάλη βελτίωση και είναι μια εγγύηση για τους εταίρους μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε χρονικούς περιορισμούς δυστυχώς, γιατί αλλιώς δεν θα τελειώσουμε την ημερήσια διάταξή μας. Κύριε ο πρέσβης του Περού, θα προσπαθώ να είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Φίσας για την παρουσίασή του. Το Περού είναι πρόθυμο να συνεισφέρει στην ολοκλήρωση του έργου του. Να κάνω μερικά σχόλια σε ό,τι αφορά την συμφωνία κατόπιν των όσων ελέγχθησαν προηγουμένως. Πρώτον, η Επιτροπή Εμπορίου που διαθέτουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που πιο καλά λειτουργεί ε, και η συμφωνία αυτή είναι αυτή που πιο, πολύ, ε, πιο πολλά ωφέλη έχει φέρει. Ποια είναι αυτά τα ωφέλη. Πρώτον, στο μην παραδοσιακό τομέα, δηλαδή διαφοροποίηση του εμπορίου μας, ε, εξαγωγές μη παραδοσιακές εξαγωγές του Περού προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν ετησίως κατά 8,3% κατά μέσο όρο. Νέες επιχειρήσεις λοιπόν, νέοι κλάδοι οι οποίοι εντάσσονται στο διεθνές εμπόριο από τη δική μας πλευρά. Είμαι πιο συγκεκριμένος. Στα πέντε χρόνια της συμφωνίας καταγράφηκαν 813 καινούρια προϊόντα τα οποία εξήχθησαν το 97,9% αυτών είναι μη παραδοσιακά προϊόντα, χημικά, μέταλλα, ε, υφάσματα. Την ίδια περίοδο 2.750 νέες επιχειρήσεις που εξάγουν ε, έλαβαν, υποφελήθηκαν τη συμφωνία. Από αυτές το 88,2% είναι μικροεπιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις. Και εδώ βλέπουμε το κοινωνικό όφελος που προέκυψε ε, από τη Συμφωνία για το Περού. 88,2% των νέων επιχειρήσεων είναι μικροεπιχειρήσεις ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μεταξύ του 2012 και του 2017 ε, η μέση αμοιβή των εργαζομένων σε ε, επιχειρήσεις που εξάγουν αυξήθηκε κατά 23,7% κατευθείαν στην τσέπη των εργαζομένων. Όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη σε, όταν κάνουμε την ανάλυση της, ε, ε, εφαρμογής συμφωνίας. Αύξηση στον αριθμό εργαζομένων. Στους μη παραδοσιακούς τομείς 3%. Στον αγροτικό τομέα και τον τροφιμικό τομέα η αύξηση έχει φτάσει το σχεδόν το 16%. 16% παραπάνω ε, οι εργαζόμενοι σε αυτόν τον κλάδο. Ο κ. Σόλτς μίλησε για την ανάγκη γεωγραφικής διαφοροποίησης των ωφελών. Να μην εντοπίζονται δηλαδή, τα ωφέλη μόνο στις μεγάλες πόλεις. Να σας πω μερικά στοιχεία. Πιούρα, Καχαμάρκα, μία από τις ε, πιο φτωχές ε, περιοχές του Περού. Λαμπαγέκη και Χουνί, όλες αυτές οι περιφέρειες, τέσσερις δηλαδή, είναι τέσσερις από τις 11 που πιο πολλά ωφέλη δέχτηκαν από τη συμφωνία. Αύξησαν τις εξαγωγές τους Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 923 εκατομμύρια, από 923 ε, εκατομμύρια ευρώ το 2012 στα, στο 1 184 εκατομμύρια το 2017 η κεντρική περιοχή του Χούνινγκ είδε τις εξαγωγές της να αυξάνονται κατά 150% εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δείχνει ότι είναι αποκεντρωμένα και τα ωφέλη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές ε, δεσμεύσεις και περιβαλλοντικές υποχρεώσεις. Ο Οργανισμό Αξιολόγησης και ε, περιβαλλοντική Φορολόγηση του Περού από το 2013 εδρεώνει μια προσέγγιση που επιτρέπει την ανάπτυξη της του, ελεύθερου επιχειρήν και να τη συνδυάζει με την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτός ο οργανισμός ε, έχει δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις, αλλά και ε, να επιβάλλει μέτρα προληπτικά και διορθωτικά. Ενημερωτικά σας λέω ότι προσφάτως το Περού ε, ενέκρινε το νόμο πλαίσιο για την κλιματική αλλαγή. Είναι το πρώτο νομοθέτημα που υιοθετείται στην περιοχή μας. Δείχνει πόσο πολύ μας ανησυχεί το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Σε ό,τι αφορά τα εργασιακά, τα οποία σχολιάστηκαν. Το Περού ε, έχει υπογράψει τις βασικές ε, συμβάσεις του, της, ε, Διεθνούς Εμπορίου. Και μάλιστα εξελέγημεν πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ILO αυτό απηχεί την αναγνώριση των προσπαθειών της χώρας μας. σε ορισμένα έγγραφα που αφορούν το Περού υποστηρίζεται, λέγονται κάποια πράγματα για τις ε, ε, επιθεωρήσεις. Οι επιθεωρητές στο Περού το 2016 ήταν 306. Φέτος το νούμερο έφτασε στους 684 επιθεωρητές εργασίας. Και ελπίζουμε ότι του χρόνου θα φτάσουν στους 855. Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα και προηγουμένω. Το άρθρο 281 του Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών δεν μα υποχρεώνει να δημιουργήσουμε ε, ένα DAC, μια ε, εσωτερική συμβουλευτική ομάδα. Θα μπορούσαμε, μπορούμε να ε, επωφεληθούμε των ομάδων που ήδη υπάρχουν. Και με αυτή, αυτή την έννοια εμείς ενισχύουμε αυτή τη συμμετοχή με πρόεδρο πλέον της ομάδας DAC ε, όχι από το κράτος, από το κράτος, αλλά εκπρόσωπο των εργαζομένων ή των εργοδοτών. Τέλος, ε, θα επαναλάβω και εγώ την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς να συμμετέχουμε σε ένα σύστημα ε, διεθνούς εμπορίου προβλέψιμο που θα βασίζεται σε ισότιμους κανόνες. Υπ' αυτή την έννοια πολλοί από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούμε α, από τη δική μας οπτική γωνία ότι θα πρέπει να την χάνουν καλύτερου συντονισμού. Βλέπω το σφυράκι στα χέρια σας, Πρόεδρε, πριν το χτυπήσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θέλετε άλλες πληροφορίες, ευχαριστώ να σας τις δώσουμε. Thanks Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρέσβη. Ένα ερώτημα είχε θέσει ο κύριος Σόλτ, μάλλον θα θέσει ένα ερώτημα, αλλά σύντομα, σας παρακαλώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομο, κύριε Πρόεδρε, γιατί θα έχουμε περισσότερο χρόνο να συζητήσουμε το σχέδιο έκθεσης όταν υποβληθεί. Αλλά αφού έχουμε εδώ πέρα και τον πρέσβη και την εκπρόσωπο της πρεσβείας από την Κολομβία, Αναφερθήκατε στην ειρηνευτική διαδικασία και γνωρίζουμε ότι έχουμε ένα νέο πρόεδρο και φαντάζομαι και μία νέα κυβέρνηση. Θα συνεχιστεί η ειρηνευτική διαδικασία. Γιατί άλλες υποσχέσεις έδωσε προεκλογικά. Πώς μπορούμε να σταθεροποιήσουμε ή να εμβαθύνουμε την ειρηνευτική διαδικασία και πώς μπορεί να συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρος, δεν είμαι σίγουρος ήταν σύντομη η ερώτησή σας. Η απάντηση τουλάχιστον δεν μπορεί να είναι σύντομη. <laughs> Ε, ε, ε, Κύριε Βάργα, έχετε το πρόβλημα. Μα... Καταχράστε το ότι είμαι γυναίκα για να μου κάνετε δύσκολες ερωτήσεις. Αλλά η απάντηση είναι απλή. Είμαστε πεπισμένοι εμείς ως πρεσβεία ότι η ρευνική διαδικασία έχει φτάσει σε όλες τις περιοχές. Είναι πλέον ανεπίστρεπτη. Εσείς ως πολιτικοί ξέρετε Άλλο είναι να κάνει κανείς ε, προεκλογική εκστρατεία και άλλο είναι να αναλάβει αξίωμα και να πρέπει να πάρει αποφάσεις. Σήμερα διάβασα ότι ο στρατηγός Ναράχο θα λάβει συγκεκριμένη εντολή να ασχοληθεί με αυτό το θέμα το οποίο δείχνει ότι η μετάβαση από την προηγούμενη κυβέρνηση στην επόμενη θα είναι ιδιαίτερα ομαλή. Είναι σημαντικό να συνεχίσετε να στηρίζετε την ειρηνευτική διαδικασία να βοηθήσετε και την ε, παρούσα κυβέρνηση ώστε η μετάβαση να είναι η ε, πιο απρόσκοπτη δυνατή. Ευχαριστώ πολύ. Η βοήθειά σας είναι θεμελιώδης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σύντομη απάντηση. Έχετε το λόγο, αλλά σύντομα, σας παρακαλώ πολύ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ είχα πολλές ε, ερωτήσεις. Δεν θα ήθελα να διαταράξω αυτή την συνετική ατμόσφαιρα που έχουμε, αλλά μήπως κρύβουμε αυτή τη στιγμή κάποια πράγματα. Η συμφωνία αυτή δεν συνάδει με τη Συμφωνία των Παρισίων. Μας είπατε ότι πρέπει να δείξουμε υπομονή εμείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά πώς μπορούμε εμείς ε, να συμβάλλουμε αυτή τη στιγμή ε, άλλα περιμέναμε από τις δικές σας τις πιστοποίησεις και από τις δικές σας τις δράσεις. Είχαμε πει ότι για τις μπανάνες, για τη ζάχαρη, για τον τομέα της αλίας είχαμε εντελώ διαφορετικές απαιτήσει. Τα όσα γράφονται αυτή τη στιγμή στην έκθεση είναι πάρα πάρα πολύ ασαφή. Επομένως, δεν μπορώ παρά να πω ότι η κατάσταση είναι δραματική για εμάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ειρηνευτική διαδικασία, ελεύθερε συναλλαγές κτλ. Πολύ ωραία όλα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως, η οποία έρχεται και μας λέει η ίδια ότι ακόμα πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, δεν μιλήσαμε καν για το σεβασμό των δικαιωμάτων στον τομέα της απασχόλησης. Κύριε Πρέσβη, ξέρετε ότι ένα 60% 17 εκατομμύρια άτομα δηλαδή εργάζονται στον άτυπο τομέα. 2,9 εκατομμύρια είναι παιδιά 6 με 17 ετών. Έκθεση του, της Διεθνούς ε, Οργάνωσης ε, Εργασίας. Και ξέρετε ότι ε, υπάρχουν πάρα πολλοί οργανισμοί, μη κυβερνητικοί οργανισμοί που λένε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προστατεύονται πραγματικά τα δικαιώματα των εργαζομένων. Και αυτό δεν γίνεται. Και ξέρετε ότι πολλές φορές είχαμε ακόμα και προσφυγή στη δικαιοσύνη και ε, μην ξεχνάμε ότι στην Κολομβία ένα 70% και το λέει αυτό ο Καναδικός Σύνολος Διεθνούς Συνεργασίας ένα 70% των εργαζομένων δεν έχουν ούτε πρόσβαση στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και πάρα πολλές από τις ε, θέσεις αυτές απασχόλησης που είναι συνήθως ορισμένου χρόνου δεν τηρούν βασικούς κανόνες αξιοπρεπούς εργασίας. Εγώ αυτή τη στιγμή νομίζω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με τους συγκεκριμένου αυτού τομεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πλήττονται και νομίζω ότι ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει να διστάζει να καταβάλει το τίμα που πρέπει να καταβληθεί κάθε φορά. Από ε, ανθρώπινης πλευράς, είτε μιλάμε για τους κατοίκους της Κολομβίας ή τους κατοίκους του Περού ή για τους κατοίκους της δικής μου της χώρας, νομίζω ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουμε, αν θέλετε, αυτή τη συμφωνία. Ήμουν αρκετά σύντομη, κύριε, κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι, προφανώς και θα επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό όταν θα υποβάλει την έκθεση του κύριο Φίσας στι 27 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα. Αλλά για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση ξαναδίνω το λόγο στον εισηγητή. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλε τι παρεμβάσει από του συναδέλφους, από διάφορε πολιτικέ ομάδε Με πολλού έχουμε συνεργαστεί και με χαρά θα ξανασυνεργαστώ μαζί τους. Συμφωνώ με την Ιμακουλάδα ε, για το ενδιαφέρον που εκφράζει και που συμμερίζομαι για τις μικρομεσαίες. Δεν υπάρχει ειδικό κεφάλαιο, άρα θα πρέπει να βρούμε ε, τον τρόπο για να τις ε, συμπεριλάβουμε. Στον κύριο Ζαχράντιλ, πολλά πρέπει να γίνουν για να βελτιωθούν οι εμπορικές συναλλαγές. Και μας ανησυχεί όλους η έλλειψη ενημέρωσης Ιδίως ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν αρκετές πληροφορίε Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κατανοήσουν τα πλεονεκτήματα προς τον ε, Helmut Scholz. Έχει δίκιο. Πρέπει να αναφέρουμε τη σύνδεση μεταξύ αυτής της συμφωνίας και της συμφωνίας ειρήνης. Το τόνισε και η εκπρόσωπος της Κολομβίας. Και βεβαίως αναγνωρίζω ότι η άτυπη εργασία εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική. Αλλά αυτό που πρέπει να δούμε είναι πού ήμασταν και πού έχουμε φτάσει. Όχι απλώς να λέμε γενικά όλα είναι άσχημα. Αυτό δεν βοηθάει. Πρέπει να δούμε σε τι κατάσταση ήταν το Περού και η Κολομβία και πού είναι τώρα. Τι προσπάθειες έχουν γίνει για βελτιωθεί η κατάσταση. Μιλήσαμε για τις εξαγωγικές εταιρείες, πόσο πολλές είναι, ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση για τα κοινωνικά δικαιώματα, για το περιβάλλον. Να μην βλέπουμε το ποτήρι μισοάδιο, να βλέπουμε ότι είναι και μισογεμάτο. Πολλά θετικά συμβαίνουν. Πασερτώσει, με χαρά θα συνεργαστώ μαζί σας. Ξέρουμε ότι για τις εκθέσεις αυτές επιτρέπονται μόνο ένας ορισμένος αριθμός λέξεων και βεβαίως θα εξετάσω και τις τροπολογίες σας να δω πώς μπορώ να τις περιλάβω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κλείσαμε με το θέμα αυτό. Αλλά θα τα ξαναπούμε στις 27 Ενάτου για να συζητήσουμε το σχέδιο έκθεσης. 11. Ad hoc ε, αποστολή στην πόλη του Μεξικού. 6-8 Ιουνίου. Είχε υπάρξει ε, καταρχήν συμφωνία για την, ε, τον εξυγχρονισμό της ε, εμπορικής συμφωνίας Ένωση Μεξικού, το οποίο ανακοινώθηκε τον Απρίλιο στην έκθεση στο Ανόβερο, στην πόλη μου, όπου συμμετείχε το Μεξικό. Σε αυτή την περίφημη εμπορική έκθεση του Ανόβερου. Η κυρία η ε, Μακουλάδα Ροντρίγκεθ Πινέριο και ο κύριος Φίσας ήταν στην αντιπροσωπεία. Να δώσω το λόγο πρώτα στην Ήμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχαριστήσω την Μεξικανική κυβέρνηση και την πρεσβεία του Μεξικού. Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την εξαιρετική υποδοχή, το εξαιρετικό πρόγραμμα εργασιών που μας προετοίμασαν και τις ευκαιρίες που μας δόθηκαν να εμβαθύνουμε σε όλα τα θέματα τα οποία μας ενδιέφεραν, που ήταν πολλά. Να ευχαριστήσω επίσης τη Γραμματεία, ιδιαίτερα την Μερθέδες Ροδρίγεθ για την εξαιρετική δουλειά που μας ε, βοήθησε πάρα πολύ στη δουλειά μας. Ε, ήταν μια αποστολή πολύ επίκαιρη προκειμένου να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα υπέρ της επικαιροποίησης της ε, Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών με το Μεξικό, ένα ισχυρό μήνυμα ε, εναντίον της πολιτικής Τραμπ, ένα κοινό μήνυμα ότι υποστηρίζουμε ένα διεθνές εμπόριο δίκαιο, ισορροπημένο που βασίζεται στον ε, διάλογο και σε κοινούς κανόνες. Όλα αυτά ήταν πολύ σημαντικά. Ο στόχος της αποστολής ήταν πρώτον να δώσουμε όλα, αυτά τα μηνύματα. Δεύτερον, να ενθαρρύνουμε το Μεξικό να προβεί στην επίλυση των εκκρεμών θεμάτων προκειμένου να ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση της συμφωνίας ιδιαίτερα στο, στην, στο άνοιγμα των δημόσιων προμηθειών στα κρατήδια του Μεξικού σε υπο επίπεδο. Η μοξικανική κυβέρνηση έχει αναλάβει αυτή τη δέσμευση έτσι και αλλιώς και επιμείναμε στην ανάγκη μέχρι το τέλος του χρόνου να ε, διαθέτουμε τον κατάλογο με, τον, με τους οργανισμούς που θα συμμετάσχουν σε αυτό το άνοιγμα των προμηθειών. Ε, μετά, να ενημερώσουμε το Μεξικό για τις βασικές μας ανησυχίες σε ό,τι αφορά την ε, υπογραφή της Σύμβασης 92 του ILO. Συναντηθήκαμε τον Υπουργό Εργασίας της Κυβέρνησης του Μεξικού και το συζητήσαμε σε βάθος. Ήδη έχουν προβεί σε μια εργασιακή μεταρρύθμιση. Η κυβέρνηση έχει υπογράψει τη σύμβαση και θα πρέπει να επικυρωθεί από τη Γερουσία. Ελπίζουμε ότι η καινούργια Γερουσία ε, όταν αλάβει τα καθήκοντά της και συσταθεί σε σώμα θα προβεί σε αυτή την επικύρωση. Συναντηθήκαμε επίσης με προσώπους της κοινωνίας των πολιτών, ε, δομημένοι από ό,τι είδαμε, Προφανώς ε, χρειάζονται περισσότερη συμμετοχή στην εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας. Νομίζω ότι οι συνθήκες υφίστανται γι' αυτό. Η βούληση υπάρχει επίσης. Ενδιαφέρουσα συνάντηση με το φορέα που σχετίζεται με τις γεωγραφικές ενδείξεις. Έχουμε και εμείς να μάθουμε πράγματα από το Μεξικό, γιατί διαθέτουν ένα φορέα, ένα οργανισμό που τους επιτρέπει να ε, επιβάλλουν ποινές αλλά να κάνουν και επιθεωρήσεις σε ό,τι αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις το ερώτημα ήταν πώς θα γίνει η συμμόρφωση μέσω της επισήμανσης ε, ιδιαίτερα για διαφορετικά προϊόντα που έχουν το ίδιο όνομα. Ε, οι δυνατότητε όμω ε, να επιβληθούν κυρώσει από αυτόν τον οργανισμό, να κλείσουν επιχειρήσεις ε, και η βεβαιότητα για την οποία μας, την οποία μας επιβεβαίωσαν ότι έχουν ότι μπορούν να συμμορφωθούν μας καθησύχασαν. Είναι ίσως ένα μοντέλο το οποίο θα μπορούσαμε και εμείς να αντιγράψουμε. σε ό,τι αφορά την ζώνη ελεύθερων συναλλαγών της Βόρειας Αμερικής, την ΝΑΦΤΑ, την ε, Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών της Βόρειας Αμερικής. Συναντήκαμε με τον Υπουργό Οικονομίας για μία ώρα πιο πολύ από ό,τι είχε προγραμματιστεί. Είχαμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας μας ενημέρωσε ότι κατά τη διάρκεια της ε, προεκλογικής εκστρατείας ε, το θέμα αυτό είχε παγώσει. Προφανώς θα πρέπει να δούμε τα τελικά αποτελέσματα. Δεν υπάρχουν πολλές ελπίδες δεδομένου ότι η Αμερικανική κυβέρνηση έχει στόχο να προωθήσει διμερείς συμφωνίες, όχι πολυμερείς όπως είναι αυτά. Ε, σπρώξαμε το θέμα του φύλου και η μεξικανική κυβέρνηση μας υποσχέθηκε ότι ε, θα ε, φροντίσει την συμπερίληψη και της πτυχής του φύλου. Τώρα, για τη γεωργία και το γεωργικό τομέα. Συναντηθήκαμε με τον Υπουργό Γεωργίας, συζητήσαμε σε βάθος επιμένουν πολύ για την ανάγκη η μεταποίηση γεωρικών προϊόντων να συμπεριληφθεί έτσι ώστε τα προϊόντα τους να έχουν μεγαλύτερη προσθέμενη αξία θα συνεργαστούν στενά μαζί μας στον συντονισμό φυτογειονομικών μέτρων το ρυθμιστικό πλαίσιο στο οποίο χρειάζεται να συνεργαστούμε περισσότερο. Υπάρχουν κάποιες ανησυχίες εκεί. Γιατί εμείς έχουμε πολύ ισχυρό κανονιστικό πλαίσιο, αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο. Τέλος, ε, νομίζω ότι η αποστολή αυτή ήταν επιτυχημένη και πάλι ευχαριστούμε τις, την κυβέρνηση και τις αρχές του Μεξικό και θέλω να επιμείνουμε στα θέματα που εκκρεμούν. Εμείς στείλαμε το μήνυμά μας ότι έχουμε την αποφασιστικότητα να κάνουμε ό,τι χρειάζεται προκειμένου η συμφωνία αυτή να ψηφιστικά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας μας. Τους είπαμε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να αρχίσει να εφαρμόζεται το συντομότερο δυνατό. Gracias. Mr. Ο κύριος Φύσης έχει το λόγο. Δεν θα προσθέσω πολλά. Μου καλά να τα είπε όλα. Ευχαριστώ τη Μερθέδες και την Επιτροπή. Και ευχαριστήσαμε, ευχαριστώ ιδιαίτερα και τον εκπρόσωπο της Ένωσης εκεί, τον Γερμανό πρέσβη που ηγείται, που μας ε, συνόδεσε παντού με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Εργαστήκαμε πολύ, οι συναντήσεις μας ήταν σε πολύ ψηλό επίπεδο. Αυτό έχει να κάνει με την καλή θέληση των συνομιλητών μας, αλλά και για το τεράστιο ενδιαφέρον που έχει το Μεξικό για να υπάρξει αυτή η συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών. Το 80% βέβαια των εμπορικών συναλλαγών του Μεξικού είναι με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Οπότε καταλαβαίνετε τι ανησυχία έχουν λόγω τη πολιτική Τραμπ. Οπότε ψάχνουν ε, νέες διεξόδους. Θέλουν περισσότερες συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα πρέπει ακριβώ να υποφεληθούμε από αυτήν την ευκαιρία. Γιατί έτσι θα ωφεληθούν και οι Μεξικανοί. Πραγματικά αυτό ε, φάνηκε και με το πόσο χρόνο διέθεσαν για μας, ο Υπουργός Εμπορίου μας δέχτηκε για πάνω από μια ώρα ε, ενώ ε, έχει πολλή δουλειά και πολλοί άλλοι υπουργοί. Και να καταλήξω με αυτό που κατέληξε και η Μακουλάδα και που με ανησυχεί πολύ. Πρέπει αυτή η συμφωνία να υπογραφεί πριν τη λήξη της παρούσης θητείας. Μου φαίνεται παράλογο ότι για λόγους μετάφρασης μπορεί να μην προλάβουμε να την υπογράψουμε. Ξέρω ότι είναι τόσο πολλές γλώσσες, παίρνει χρόνο η μετάφραση, 24 γλώσσες, πρέπει να την εγκρίνουν μετά και οι νομομαθείς, ε, οι γλωσσομαθείς ε, νομικοί, αλλά είναι πιο περίπλοκη η μετάφραση από την ίδια την ε, διαπραγμάτευση της συμφωνίας. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Πρέπει να προλάβουμε να ψηφίσει και η Ολομέλεια πριν το τέλος της θητείας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. παρακαλώ. Νομίζω ότι το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον άκουσα τον απολογισμό αυτό της επίσκεψης από τους δύο συναδέλφους. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι στο Μεξικό έχουμε προεδρικές εκλογές την 1η Ιουλίου. Και βέβαια ξέρετε ότι οι δημοσκοπήσεις μπορούν να κάνουν λάθος. Λένε ότι ο κύριος Σομπραντόρα από την αριστερά θα εκλεγεί. Και ο κύριος Σομπραντόρα, από ό,τι φαίνεται, είναι σαφώς κατά των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών και γενικά κατά της παγκοσμιοποίησης. Και αυτό δεν αναφέρθηκε καν από τους συναδέλφους. και βλέπω τον συμπαθέστατο συνάδελφο να γνέφει αυτή τη στιγμή, θα μπορούσε τουλάχιστον να το έχει αναφέρει αυτό. Το ότι έρχεστε εδώ πέρα και αναφέρεστε κατά αυτόν τον τρόπο στην επανακύρωση της συμφωνίας αυτής, ενώ μπορεί να καταργηθεί από τη μία μέρα στην άλλη, δηλαδή σε τρει μήνε μετά την 1η Ιουλίου μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Το ότι δεν κάνετε καμία αναφορά σε αυτό μου φαίνεται πραγματικά περίεργο. Γνωρίζουμε τι πρεσβεύει ο κύριο Μπρεντόρ. Έχω διαβάσει βέβαια άρθρα στον τύπο κυρίω, αλλά έχουμε και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει μια πολύ σημαντική αντιπροσωπεία στο Μεξικό. Θα έπρεπε ίσω αυτοί να μα ενημερώσουν περί τίνο πρόκειται είναι υπερβολικές αναφορές αυτές. Πρόκειται όντως ο κύριος Ομπραντόρ να καταργήσει αυτή τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Τι θα γίνει στην πράξη. Δεν μας αφορά καθόλου τελικά η οι εκλογές αυτές είναι τελώς ουδέτερε από πολιτικής πλευράς. Θα πρέπει να με ανησυχούν ενδεχομένως αυτές οι εκλογές. Πραγματικά θα ήθελα να μάθω από τους συναδέλφου. Ήρθα εδώ, περιέργοζα μια φορά, για να ακούσω και να μάθω από τους συναδέλφους. Ο κύριος φίσα έχει το λόγο. Αγαπητέ συνάδελφε Λόρδε Ντάρτμουθ, δεν θα αποφασίσω εγώ τι θα πει ένας αριστερός πρόεδρος. Η πολιτική στο Μεξικό είναι διαφορετική από την πολιτική στην Ευρώπη. Πολλές φορές οι αντιπαραθέσεις είναι πολύ έντονες και ε, απροσδόκητες από τις επαφές που είχαμε. Και εγώ εξεπλάγιν. Νόμιζα ότι είναι έξαλλος ε, αριστεριστής ο Ομπραδόρο, όπως μας τον περιέγραφαν, αλλά φαίνεται ότι αλλάζει τώρα. Και οι συνεργάτες του είπαν ότι θα, θα σεβαστούν πλήρως τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών. Δεν εξέφρασαν καμία επιφύλαξη. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε τι έκανε ο κύριος Ομπραδόρ όταν ήταν δήμαρχος του Μεξικού που δεν είναι και κανένα χωριουδάκι και ήταν πολύ επιτυχημένος. Το κόμμα που είναι πιο κοντά στο δικό μου κόμμα, το κόμμα ΠΑΝ, Υπάρχουν δύο πρώην πρόεδροι του ΠΑΝ που στηρίζουν τον κύριο Ομπραδόρ και 32 προσωπικότητες του ΠΑΝ αυτή τη στιγμή κατεβαίνουν ε, για δήμαρχοι, για γερουσιαστές ε, με αυτή την ομάδα που λέγεται Μορένα. Δεν ξέρω αν μπορεί να θεωρηθεί ότι για λόγους καιροσκοπικούς έχουν αλλάξει άποψη. Αλλά από ό,τι μου είπαν, ο Λόπεθ Ομπραδόρ είναι ιδιαίτερα ρεαλιστής και με αυτό μας το είπαν όχι μόνο οι δικοί του, αλλά και ο πρέσβης της Ένωσης και οι άλλοι πρέσβεις ε, χωρών της Ένωσης με τους οποίους συναντηθήκαμε. Και ασχολείται ιδιαίτερα με το θέμα αυτό. Ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να εάν δεν εγκριθεί μέχρι τη λήξη της θητείας και περιμένουμε να εγκριθούν και οι δικοί μας επίτροποι και η δική του ομάδα θα πρέπει να περιμένουμε να εγκριθεί αυτή η συμφωνία μέχρι το 2020. Γι' αυτό είναι σημαντικό να επιχειρήσουμε να επιταχύνουμε όσο γίνεται. Ευχαριστώ τον κύριο Ντάρτμουθ που έκανε αυτή την παρατήρηση. Έπρεπε και εγώ να το είχα σχολιάσει. Πράγματι, κατά τη διάρκεια της αποστολής μας διαπιστώσαμε την ομόφωνη υποστήριξη όλων και των πολιτικών κομμάτων και της σημερινής κυβέρνησης και της κυβέρνη... κοινωνίας των πολιτών. Όλοι υποστηρίζουν την Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών. Συναντήκαμε και με όλους τους πρέσβεις των κρατών μελών στο Μεξικό και μας υπεβεβαίωσαν ακριβώς το ίδιο όλοι οι υποψήφοι υποστηρίζουν τη συμφωνία, οπότε ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών, η συμφωνία δεν κινδυνεύει. Όλοι είναι υπέρ της εμβάθυνσης των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να επιτύχουμε τη σύναψη αυτή, την επικαιροποίηση στο στομότερο δυνατό, προχωρήσουμε γρήγορα και με τις μεταφράσεις, ας γίνει ο ενδελεχής νομικός έλεγχος. Λοιπόν, καλή τύχη και καλή δύναμη σας εύχομαι. Ολοκληρώνεται αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης και περνάμε στο τελευταίο για σήμερα, το σημείο 12. όπου έχουμε τη Συμφωνία Συνεργασία για την Εταιρική Σχέση και την Ανάπτυξη μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ισλαμική Δημοκρατία του Αφγανιστάν. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία τροπολογία για την έκθεση που θα συντάξει η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Και αυτό διότι στην συμφωνία αυτή συνεργασία για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ισλαμική Δημοκρατία του Αφγανιστάν καλύπτονται και εμπορικά ζητήματα. Το πρόβλημα τώρα όμως είναι περισσότερο θεσμικής φύσης, διότι μετά την υπογραφή της 18 Φεβρουαρίου 2017 άρχισε να ισχύει προσωρινά το συμβούλιο, ήδη, το, συγγνώμη, η συμφωνία αυτή ήδη από την 1η Δεκεμβρίου, χωρίς να υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο εμείς υποβάλαμε μια τροπολογία στην έκθεση της Επιτροπής ΑΦΕΤ, λέγοντας ότι σε καμία περίπτωση αυτό δεν συνάδει μετά όσα προβλέπει η συνθήκη. Και γι' αυτό το λόγο κάνουμε μια σαφή δήλωση, σε αυτή την τροπολογία, λέγοντας ότι θα πρέπει να τηρηθούν και οι διαπραγματεύσεις μας με το Συμβούλιο στα πλαίσια της διοργανικής συμφωνίας, όπου λέγεται ξεκάθαρα ότι δεν θα πρέπει να έχουμε προσωρινή εφαρμογή συμφωνιών αν δεν έχει δοθεί πρώτα η σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκτός και αν συντρέχουν εύλογοι λόγοι, όπως για παράδειγμα επίγουσες καταστάσεις. Εδώ όμως άρχισε να ισχύει μετά από έξι μήνες, δεν υπάρχει κάτι το επίγον Λοιπόν, θα ήθελε από αυτού να πάρει κάποιο το λόγο. Ουδής. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ενδεχομένως θα ήθελε να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ως Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση εκτιμούμε ιδιαίτερα την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτή τη Συμφωνία συνεργασία για την Εταιρική Σχέση και την Ανάπτυξη μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Αφγανιστάν. Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα προκειμένου να βαθμιστεί η σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση και Αφγανιστάν και προκειμένου να έχουμε μια στρατηγική ευρωπαϊκή απέναντι στο Αφγανιστάν. Η εφαρμογή τώρα τη συμφωνία αυτή, η προσωρινή τη εφαρμογή, είναι πάρα πολύ σημαντική προκειμένου να πετύχουμε αυτό το στόχο. Θα καταφέρουμε να αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε περισσότερο σε τομείς αρμοδιότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης μία ώρα αρχίτερα ουσιαστικά. Και όντω υπάρχει ένα κλάδο που έχει να κάνει με εμπόριο και με επενδύσει. Αλλά το κεφάλαιο αυτό έχει να κάνει ουσιαστικά με συνεργασία, με ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά ζητήματα εμπορικά και επενδυτικά. Δεν έχει να κάνει με πρόσβαση στι αγορά, δεν έχει να κάνει με απελευθέρωση των συναλλαγών. Συνεπώς, εφόσον δεν είναι συμφωνία σύνδεσης, αυτή η συμφωνία συνεργασίας δεν περιλαμβάνει ουσιαστικά, αν θέλετε, ένα mini FTA, μια μικρή συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, μα νομίζω ότι εδώ διαφωνούμε. Επί της αρχής διαφωνούμε. Θεωρώ ότι και στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας, που όπως είπατε είναι συμφωνία εταιρικής σχέσης και ανάπτυξης, δεν θα πρέπει να προβλέπεται εξαίρεση. Δεν θα πρέπει δηλαδή να αρχίσει να ισχύει προσωρινά αυτή η συμφωνία αν το Κοινοβούλιο δεν έχει δώσει τη σύμφωνη γνώμη του. Ακόμα στη φάση διαπραγμάτευση είμαστε με αυτή τη συμφωνία. Είπα ότι εκπροσωπή ω Μογκερίνε έκανε μια συμβαστική πρόταση προς το Συμβούλιο. Αξιολογήστε τη λίγο και αυτήν. Αλλά πέρα από αυτό, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να υιοθετήσουμε την προτινόμενη αυτή τροπολογία αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε το τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο το πρωί